good morning everyone. We Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να μιλήσω την μητρική μου, δηλαδή τα γερμανικά. Στην προ... τελευταία δημόσια κρόαση μας ε, και σήμερα το πρωί λοιπόν σε 2,5 ώρες θα ασχοληθούμε με το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος και το θέμα της NLB της ε, Σλοβενικής εταιρεία ε, και τις ε, σχετικές αποκαλύψεις. Στο πρώτο λοιπόν πάνελ έχουμε την περίπτωση του Χνοτικού Ομίλου Σλοβενία και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι έχουμε 15 γλώσσες, δερμηνία σε 15 γλώσσες Ευχαριστούμε τους ερμηνείς. Και έτσι έχουμε και web streaming αυτή τη φορά. Έχουμε και μια ελαφριά καθυστέρηση. Δεν θέλω λοιπόν να μακρηγορήσω εισαγωγικά. Η σημερινή ακρόαση στο πρώτο τμήμα τη θα κοιτάξουμε την, ε, το χρησιμοποιητικό όμιλο NLB και τις ε, σχετικές ε, αποκάλυψεις και στα δεύτερο του σκέλος σήμερα το απόγευμα της Αγκρόση, θα δούμε ε, τα έγγραφα Paradise και των υπόλοιπων ε, επιπτώσεων. Καλώς ορίζω λοιπόν δύο ομιλητέ ομιλητές για την περίπτωση αυτή τη NLB Σλοβένια, Σλοβενίας, ε. ένα μέλος του Σλοβενικού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής που ασχολείται με τις ε, υποθέσεις αυτές και ύστερα από την ε, εφημερίδα Κότμη Ματίνα ε, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε όλους τους ομιλητές. Έχουμε 7 λεπτά για τον καθένα. Στην συνέχεια θα έχουμε τις ερωταπαντήσεις από τους συναδέλφους και έχουμε οργανώσει λοιπόν την των ερωταπαντήσεων ένα λεπτό. Οι ερωτήσεις τρία λεπτά, οι απαντήσεις προκειμένου να μπορούμε να έχουμε χρόνο. Και τώρα να δώσω τον πρόεδρο της Επιτροπής του Σλοβανικού Κοινοβουλίου α, το λόγο. Κύριε Λούκα, έχετε λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον λοιπόν θέμα. Ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει μια κάποια έκπληξη σε κάθε περίπτωση. Είχα, και μια προτιμα... Είχα προετοιμάσει και μια παρουσίαση. Θα σας παρακαλώσω λοιπόν να προχωρήσετε στις διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε λοιπόν μια σύντομη περιγραφή τι ορίζεται ως ε, άμα ξέπλυμα βρωμικού χρήματος και ποιες είναι οι υπούτες αυτές Οι τρεις φάσεις της διαδικασίας βλέπετε ποιες είναι αυτές. Σε ό,τι αφορά μια κρατική τράπεζα. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2006 στις Παρθένες νήσους με 2 δολάρια Αμα, καταστατικό κεφάλαιο. Η εταιρεία αυτή σταμάτησε να λειτουργεί, στάλτηκε τη στερεότητά του ε, το 2007 λόγω ε, υποπτών δραστηριοτήτων. Επρόκειτο λοιπόν για μια εταιρεία που είχε λογαριασμού σε δύο τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τραπεζών. με τις οποίες απαγορεύουν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΑΕ να γίνουν δια... συναλλαγές γιατί είναι ύποπτες. σε ό,τι αφορά την ε, τράπεζα Export Development Bank of Iran, του Ιράν. Η τράπεζα αυτή προστάθηκε το 2010 στον κατάλογο και με την εταιρεία λοιπόν αυτή δεν επιτρέπονται συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για το την χρηματοπιστωτική δομή της εταιρεία αυτής. Όλες οι εταιρείε που έχουν ιδρυθεί εντός ε, δύο χρόνων έχουν ε, μεταφέρει ένα δις ε, ε, δολάρια στην NLB, η οποία, όπως σας είπα, έχει ιδρυθεί με ιδρυτικό κεφάλαιο 2 δολάρια. Και συνεχίζω. Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξή. Μία ημέρα ε, μεταφέρθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε 50 μικρότερες συναλλαγές και έτσι μέχρι 70 εκατομμύρια ευρώ ε, μεταφέρθηκαν από την NLB μέσα σε δύο χρόνια. Ένα δις δολάρια σύνολο. Το 2008 η εταιρεία Φάρακ με δικό κεφάλαιο επίσης δύο δολάρια κατέστησε ο μεγαλύτερος πελάτης του NLB. Μεγαλύτερη και από έναν φαρμακευτικό γίγαντα, ο οποίος ε, είχε συναλλαγές με τη Ρωσία. Το 2009 λοιπόν, οι απασχολούμενοι, οι υπάλληλοι της τράπεζας, επεσήμεναν ύποπτες συναλλαγές και ενημέρωσαν τους, ε, τους ε, προϊστάμενους του Ωστόσο, η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί, λες και δεν είχαν απαγγελθεί, δεν είχαν επισημανθεί αυτές οι ύποπτες συναλλαγές. Το Μάρτιο του 2010, αλλοδαπές ε, συναλλαγές ε, εντοπίστηκαν, οι οποίες θεωρήθηκαν ε, ύποπτες η Γαλλία λοιπόν απέφτεινε δύο αιτήματα διευκρινήσει και η απάντηση ήταν ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι υποπτέ συναλλαγέ. Παρακαλώ λογίστε τι υποψίε σα και στη συνέχεια ε, υπήρξαν άλλες δύο καταγγελίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από χώρε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή ξεκίνησε από τις σλοβενικές αρχές ε, έρευνα, αλλά οι συναλλαγές συνέχισαν εξεγάγονται χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα πρόσκομα. Και όταν ξεκίνησαν έρευνε από την αρμόδια Σλοβενική Αρχή, τα χρήματα εξακολουθούσαν να μεταφέρονται σε λογαριασμού στην Ευρώπη, στην Αμερική και το καθεξής μέχρι τα τέλη του 2007. Το 2011 η αστυνομία ερεύνησε τις περιπτώσεις αυτές, τις υποθέσεις αυτές και όταν άλλαξε η κυβέρνηση σε δύο μήνες μόλις η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε εκκρεμής, από ανοιχτή εκκρεμής. Αυτές είναι δηλαδή οι υποθέσεις οι οποίες παραμένουν ανοιχτές, αλλά δεν ε, ερευνώνται πλέον. Παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία δεν είχε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Ήταν ενημερωμένοι βέβαια οι πολιτικοί παράγοντε, αλλά δεν υπήρχε κάποιο συμπέρασμα. Ούτε στην καινούργια NLB άλλαξε κάτι. Στη συνέχεια αναστέλησαν οι συναλλαγέ και οι δραστηριότητε με την τράπεζα Φαρούκ, αλλά όχι λόγω του νόμου. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω μόνο τα όσα διαπιστώσαμε στην έκθεση της ερευνητική Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο και ανακαλύψαμε λοιπόν ότι οι αρμόδιοι ενημερώθηκαν μεν, αλλά δεν ανέλαβαν δράση. Η διεύθυνση της τράπεζας δεν έδρασε και δεν αντέδρασε καθόλου, παρά το γεγονός ότι ήταν ενημεροί. Και η τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια δεν κινητοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα εντοπισμού α, υποθέσεων ξεπλήματος χρήματος. Και ζητήσαμε λοιπόν από την ε, δίωξη και από την αστυνομία να ερευνήσει αυτές τις υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον συνάδελφο. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία καταδεικνύει ότι από μια μικρή επιχείρηση μπορεί να γίνει μεγάλο ξεπλήμα χρήματος. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Μπορμακίνα, τον δημοσιογράφο που ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά. Ah. Okay. Uh, σας ευχαριστώ. Είμαι από την εφημερίδα Μλάντινα. Κάναμε έρευνε γύρω από την υπόθεση της NLB. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας να σας παρουσιάσω το πλαίσιο της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης για να κατανοήσετε λίγο το πώς λειτουργήσε. Στην πρώτη διαφάνεια δεν βλέπετε, αλλά αυτό το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε είναι το διεθνές πλαίσιο γύρω από την υπόθεση αυτή. Αριστερά βλέπετε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Στη μέση ε, στη μεσαία στήλη θα δείτε ε, χρήματα τα οποία uh, uh, uh, χρήματα λοιπόν τα οποία προσπορίστηκαν παρανόμως αυτοί που τα εκμεταλλεύθηκαν αλλά βλέπουμε ότι και μεγάλες τράπεζες όπως η BNP Paribas έκαναν διάφορες συναλλαγές με 190 δις. Η Commerce Bank 253 δις που είναι και το απότατο όριο αν θέλετε. Στην ουσία την τελευταία δεκαετία όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν συναλλαγές με το Ιράν. Κάποιες από τις συναλλαγές αυτές είναι πραγματικά τεράστιες από τεράστιες τράπεζες με μεγάλη ιστορία. Δεν υπήρξαν ποινικέ συνέπειε σε μια πρώτη φάση, αλλά από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ε, υπήρξε ένα πρόστιμο που ξεπέρασε τα 8,9 δις δολάρια. Βλέπετε λοιπόν ότι όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξέπλυναν πάρα πολύ χρήμα και ε, πήραν πρόστιμα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Τι έκαναν, η Commerzbank σαν παράδειγμα είχε μια ομάδα υπαλλήλων η οποία συνέλεγε τις λεπτομέρειες και τα προσωπικά, ή μάλλον διέγραφε τα προσωπικά στοιχεία των Ιρανών ε, μετά από τις συναλλαγές τις οποίες έκαναν οι Ιρανοί πολίτες. Αν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας περισσότερο στην γαλλική περίπτωση θα δούμε ότι στη 31 Μαΐου του 2014 η, Ευρωπα... Γαλλική Κεντρική Τράπεζα είπε ότι η ΜΠΕ ε, το κάνει μεν αυτό αλλά δεν παραβιάζει κάποιο ευρωπαϊκό ή ε, γαλλικό νόμο. Και ο Γάλλος Υπουργός ε, Εξωτερικών είπε ότι είναι παράλογες και μονομερείς οι επιβολές προστήμων από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πρόστιμα αυτά επιβλήθηκαν στα πλαίσια με εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω ότι λόγω όλων αυτών των γεγονότων οι ευρωπαϊκές τράπεζες φοβούνται ε, για τις υποθέσεις αυτές ακόμα. Έφυγαν φυσικά, εγκατέλειψαν το Ιράν. Είναι, δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο θα ασχοληθούν το Ιράν ξανά. το βασικό που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι στην περίπτωση του Ιράν υπήρξε μια διεθνής διαφορά ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις κυρώσεις και με τις σχέσεις με την Μέση Ανατολή. Στην Σλοβενία μία κυρία, η υπάλληλος της NLB, ήταν υπεύθυνη και έπαιρνε τις αποφάσεις για τέτοιου είδους θέματα. Όταν οι Ιρανοί πολίτες ερχόντουσαν στις τράπεζές μας στη Σλοβενία, ήταν δική της ευθύνη να παίρνει αποφάσεις για τις συναλλαγές τους. Υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετώπιζαν την υπόθεση αυτή. Λοιπόν τώρα οι εξηγήσει οι οποίες δόθηκαν γιατί δηλαδή οι Ιρανοί πολίτες είχαν έρθει στην Σλοβενία ενώ στο παρελθόν τις συναλλαγές τους τις έκαναν στην Ελβετία. Η απάντηση είναι απλή, είναι λογική. Η NLB δεν έχει ε, παράρτημα στις Ηνωμένε Πολιτείες και δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις Ηνωμένε Πολιτείες. από την εποχή της Ιουκοσλαβίας ήταν σε ένα δίκτυο τραπεζών με συνειλεγματικές συναλλαγές υψηλό ε, ποσοτικού επίπεδου και από το 2008 υπήρξαν ε, διαφορετικές ρυθμίσεις νομικές ε, για το συνάλλαγμα σε δολάρια τουλάχιστον στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ίσχυσε και για την LNB. Ήταν σαν να ήξεραν όλοι ότι μιλάμε για ξέοπλη παυρώμικου χρήματος, εκτός από την κυρία που έπαιρνε τις αποφάσεις στο NLB. Όπως είπαμε το 2008 ήρθαν κάποιοι Ιρανοί πολίτες είχαν συστατικές επιστολές από την Credit Suisse. Το Φλεβάρι του 9 έγιναν οι πρώτες συναλλαγές. ...890 εκατομμύρια ευρώ πέρασαν από τις συναλλαγές αυτές, ξεπλήθηκαν από τις συναλλαγές αυτές τα χρήματα πήγαν στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και πολλές φορές επέστρεψαν και από άλλες μεγάλες τράπεζες όπως 30 εκατομμύρια από τη Standard Checkered Bank του Ντουμπάι Λοιπόν, το 9 και το 10 υπήρξε πραγματικά μια χιονοστιβάδα αντιδράσεων γιατί οι γαλλικές αρχές άρχισαν να θέτουν ερωτηματικά για κάποιες από τις συναλλαγές αυτές και γι' αυτό τέθηκε και σε λειτουργία επιτέλους και ο εσωτερικός μηχανισμός της Σλοβενίας σε συνεργασία με τις ομάδες επιθεώρησης της Κεντρικής Σλοβενικής Τράπεζας, τις αστυνομικές αρχές δίωξης οικονομικού εγκλήματος, ε, Αυτά τα οποία λοιπόν βρήκαν ήταν ότι υπήρχαν δύο παράνομες συναλλαγές στις οποίες συμμετείχε η Iran Export Bank συνολικά 360.000 ευρώ γιατί εκείνη την εποχή στην LNB ελέγχαν όχι με υπολογιστές αλλά με το χέρι για το πώς γίνονταν οι συναλλαγές αυτές και φαίνεται ότι ξέφυγε από την προσοχή της υπεύθυνη υπαλλήλου η συναλλαγή αυτή ή μάλλον οι δύο συναλλαγές αυτές. Στο τέλος έγιναν κάποιες εσωτερικές αλλαγές στην LNB και ε, έθεσε σε λειτουργία και το καινούριο σύστημα πληροφορικής, το Siron IML Robot, το οποίο μπορεί να ελέγχει ακριβώς και τις πολλαπλές προελεύσεις κάποιων ποσών, τα οποία κατατίθενται έστω και προσωρινά στην τράπεζα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια τυπική διαφορά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα επιβολής κυρώσεων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περίπτωση του Ιράν. Ήρθε στην επικαιρότητα η αδυναμία που έχουν οι κεντρικές τράπεζες να ελέγξουν τις συναλλαγές αυτές και η υπόθεση αυτή είναι πολύ γνωστή στην Σλοβενία λόγω και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Φυσικά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Σλοβενία στον τομέα της, των φορολογικών παραδείσων. Ευχαριστώ κύριε Μακίνα για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Και για τις ε, δύο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Έχουμε τους δύο συγκητές μας. Ε. Και επειδή έχει περάσει και η ώρα, θα σας παρακαλούσα να μιλήσετε δύο-τρία λεπτά αντί για πέντε. Ο συγκητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί υπάρχει πίεση χρόνου. Πρώτα απ' όλα, μία ερώτηση προς τον ε, κύριο Λόγκαρ και τον κύριο Μαγκίνα επίσης. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η αστυνομία και οι δικαστές στην Σλοβενία ε, τι ακριβώς έχουν πράξει ως τώρα για τη δίωξη όσων εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις νομιμοποίησης ξεπλήματος χρήματος. Και αν δεν έχουν αναλάβει δράση, ποιος είναι ο λόγος. Δεύτερον, όπως είπατε κύριε Μεκίνα, είναι μια υπόθεση ευρωπαϊκή και διεθνής που αφορά περισσότερες από μία τράπεζα, σε περισσότερες από μία χώρες. Ίσως, όπως συζητήσαμε στην Επιτροπή, θα διευκόλυνε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές όπως την Europol κάτι ανάλογο έστω για να υπάρχει επιβολή του νόμου και ανάλογη κριτική δράση και εντό Ευρώπη και εκτός για να μπορούν να ερευνήσουν τέτοιες υποθέσεις και να αποκαταστήσουν ε, το νόμο, το δίκαιο στη Σλοβενία και αλλού. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, εσεί πρώτο, ό,τι αφορά και τις ε, ποιε θα είναι οι συνέπειες των όσων αποφάσισε για το Σλοβενικό Κοινοβούλιο. Πείτε. Για το ε, θέμα τη δικαιοσύνη, η εισαγγελία δεν ενημερώθηκε και γι' αυτό δεν μπόρεσε να αναλάβει και δράση. Σε ό,τι αφορά την αστυνομία τώρα, η ο υπεύθυνο έπεσε από μια σκάλα ο υπεύθυνο τη αστυνομική έρευνα έχασε τη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι η δίωξη αυτού του εγκλήματο ε, γίνεται από τον ίδιο αστυνομικό υπεύθυνο, ο οποίος διατείνεται ότι όλα ήταν εντάξει. Ο πτέος, βοηθός ε, και νυν επικεφαλής ε, της Εθνικής υπηρεσίας δίωξης. Ο πρώην επικεφαλής της δίωξης είναι πλέον επικεφαλής της εγγελίας. Όλοι δηλαδή οι ευλεκόμενοι τελικά προήχθηκαν σε πιο υψηλή θέση. Αυτό είναι προφανώς και ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Η Ερευνητική Επιτροπή, δε, απέτησε να γίνουν σχετικά βήματα. Η αστυνομία ενέργησε, εντόπισε υπό τις διαδικασίες και αναζήτησε και στους κόλπους της αστυνομίας. Τι γινόταν. Ε, και μια ειδική ομάδα για την έρευνα των αξιόπινων πράξεων, οι οποίες δεν ερευνηθήκαν από την αστυνομία. Εντοπίστηκαν λοιπόν με τον τρόπο αυτό που πολλέ τέτοιε δραστηριότητε ή υποπτέ. Για αυτά που είπε τώρα ο κύριο Μεκίνα, θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Πολλά από αυτά που λέτε δεν ε, στέκουν. Αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της τράπεζας Τη διεύθυνση τη τράπεζα εντόπισαν και ενημέρωσαν για τι ατασταλίες, αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο. Μέσα στη διάρκεια κάποιων μηνών, ε, και θα σας περιγράψω τη διαδικασία του τι έγινε, μέσα σε, διά, σε κάποιους μήνες, 22 φορεί ε, για την αντιμετώπιση ξεπλήματο βρώμικου χρήματο στον κόσμο ε, ενημερώθηκαν για την υπόθεση. Επίσης, η σχετική κοινότητα που συγκεντρώνει πληροφορίες, μυστικέ πληροφορίες για τα θέματα αυτά, ε, από άλλες χώρε βεβαίως, η έρευνα δεν οδήγησε σε κάποιο συμπέρασμα. Οπότε οι διάφορες χώρες δεν είχαν χειροπιαστά αποδεκτικά στοιχεία. Αλλά με την αναδιάρθρωση της εσωτερικής τράπεζας, την εσωτερική αναδιάρθρωση της τράπεζας NLB βρέθηκαν τα σφάλματα, ελέγχθηκε ο κατάλογος κυρώσεων ε, στις τράπεζες και αναβαθμίστηκε το σύστημα της τράπεζας. Σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύστημα για την άλλη σας ερώτηση δηλαδή, νομίζω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σας έχει απασχολήσει το θέμα του κατά πόσον πρέπει να επαναφερθούν κυρώσεις στο Ιράν και αν θα αντιταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι σε αυτήν την απόφαση. Έχετε δημοσιεύσει και πολλά κείμενα ε, προς τις τράπεζες ε, για να γίνουν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες λίγο σαφέστερες. Δηλαδή οι συναλλαγές που έχουν με το Ιράν. Το πρόβλημα όμως που παραμένει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξωεδαφικές δυνατότητες και μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε τράπεζες Ναι, ο, ο κύριος ε, Λουγκάρ. Να σας πω ότι ενημερώθηκαν 33 υπηρεσίες μεν. Αλλά η δική μας υπηρεσία δεν ε, ε, μίλησαν, δεν ανέφεραν 680 εκατομμύρια, αλλά 680 χιλιάδες ε, δολάρια. Αυτή είναι η διαφορά και να σας πω ότι ε, δεν ενημερώθηκε ούτε οι σχετικές μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, ούτε τον ΙΠΑ. Πρόκειται για μια επιλεκτική τέτοια καταμέτρηση. Γιατί, δεν ξέρω, ε, καταλήξουμε, καταλήξαμε σε λάθη σε ό,τι αφορά το συνολικό πόσο, γιατί γίνεται αναφορά για 680 εκατομμύρια και όχι 680 χιλιάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαι σύντομος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τι έκανε ο Ελβετικός Φορέας για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Με τη συναλλαγή με τη Σλοβενία είπαν με πολύ κοινικό τρόπο ότι κάθε ε, συναλλαγή από, την, από το εξωτερικό δεν μπορεί να θεωρηθεί ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με πολλή ηρωνία. Ευχαριστούμε ο κύριος Γιάτσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριοι για τις παρεμβάσεις σας. Διερωτώ με κατά πόσον τέτοιε εγκληματικέ δραστηριότητε, τέτοια κλίμακα σε αυτό το τομέα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει νέα νομοθεσία που ισχύει, υπάρχει νέα νομοθεσία υπό εξέταση και έγκριση αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την περίοδο που ξεκίνησαν όλα αυτά και το σήμερα, όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά, υποθέτουμε, ως προς την εντοπισμό τέτοιων δραστηριοτήτων. Εξ όσων γνωρίζω, αποφασίστηκε να καταγράφονται οι δικαιούχοι των εταιριών ε, και των ομίλων και οι πληροφορίες των δικαιούχων των ιδιοκτητών να είναι γνωστές στο κοινό η ανάληψη μέτρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ε, έχουμε, ε, έχει, ελπίζουμε, θα έχει, ελπίζουμε, τη δυνατότητα να εμποδίσει τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Μεκίνα. Ναι, τα στατιστικά στοιχεία που έχω εγώ να εξηγούν, αυτό ήταν ένα τυχές ε, συμβάν βεβαίω. Αλλά βάσει τη έκθεση τη Τράπεζα τη Σλοβενία για το 2014, είπαν ότι οι νέες πρακτικές της τράπεζας NLB θα έχουν ως εξής. Διότι όπως προείπα, η τράπεζα αυτή έχει ένα νέο σύστημα υπολογιστών με ρομποτικό έλεγχο όλων των συναλλαγών. Το 2014 το σύστημα αυτό επέτρεψε στον φορέα της Σλοβενίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος να έχει κατά 74% επιτυχία ανείχνευση υποθέσεων. Δεν μιλάμε για την αυτόματη ε, υποβολή εκθέσεων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, αλλά μιλάμε για τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών από πραγματικού ανθρώπου, πραγματικού υπαλλήλου στο σχετικό φορέα. Το 74% των υποθέσεων που είχαν εντοπίσει λοιπόν οι υπολογιστέ ελέγχθηκαν ε, και ήταν ε, υποθέσει που έπρεπε να ερευνηθούν περαιτέρω. Πιστεύω λοιπόν ότι το σύστημα πλέον λειτουργεί. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ και με εκπλήσουν οι δηλώσει του συναδέλφου Μακίνα. Μιλάω ω εκπρόσωπο πειράρ της Νόβλα Λιουμπλιάνσκα Μπάνκα, η οποία πριν από κάποιο καιρό ήταν συνειδιοκτήτρια μιας εταιρεία στην οποία ανήκει και η εφημερίδα Μλαντίνα. Οι χρηστές δημοσιογραφικές πρακτικές ωστόσο δεν συνεπάγονται να δικαιολογούμε κακές πρακτικές στις τράπεζες για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για μια εγκληματική διαδικασία, για μια εγκληματική ενέργεια η οποία θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και είναι πραγματικά κρίμα που η πολιτική καλείται να ερευνήσει κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσει η δημοσιογραφία, ο δημοσιογραφικός κόσμος. Σήμερα έχει αλλάξει η νομοθεσία για το τραπεζικό κλάδο για την αποτροπή τέτοιων περιπτώσεων ε, ξεπλήματος ε, χρήματος και η Νόβα Λουμπλιάνσκα Μπάνκα μέχρι το 2012 δεν είχε κανέναν έλεγχο σε ό,τι αφορά την αποτροπή ξεπλήματος ε, βρωμικού χρήματος. Η Τράπεζα της Σλοβενίας δεν παρενέβησε επίσης και προφανώς θα πρέπει να θεωρηθεί ότι φέρει ένα κόμμα τη ευθύνη όλες οι μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλήματος δρόμικου χρήματος παρουσιάστηκαν πριν από το 2007. Στη συνέχεια άλλαξε το τραπεζικό σύστημα. Οποιοδήποτε είχε κακές προθέσεις, αναγκαστικά θα πρέπει να ψάξει μια άλλη τράπεζα. Και έτσι λοιπόν αναμορφώθηκε ο κλάδος ατυχώς στην Σλοβενία ο πρόεδρος. Να κάνω μια γενική παρατήρηση Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, σύμφωνοι, αλλά εδώ θα θέλαμε να διευκάνουμε τι γίνεται. Έχετε το λόγο, κύριε Μεκίνα. Απλώς να προσθέσω σε σχέση με τις κατηγορίες. Σε σχέση με το δημοσιογραφικό έργο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έστειλα χθε. Μάλλον, σα έστειλα μια επιστολή σε όλου σα, γιατί χθε λάβατε μια τυχή επιστολή. Σα έστειλα ένα email, λοιπόν, και επειδή ε, παρέθεσα στοιχεία από την έκθεση τη Τράπεζα τη Σλοβενία, όχι τη Τράπεζα NLB. Ε, και το τρίτο που έχω να πω είναι ότι δεν ε, υπερασπιζόμαστε εδώ την Τράπεζα NLB. Η θέση μα είναι ότι αυτή δεν είναι η σημαντικότερη υπόθεση ε, συναλλαγών offshore στη Σλοβενία. Η Σλοβενία έχει προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Ρωμάνα Τόμψ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Και θα ήθελα να θέσω όλη αυτή την ιστορία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αν μου επιτρέπετε, γιατί θα καταστεί με τον τρόπο αυτό σαφέστερα και για τους συναδέλφους. Η τράπεζα για την οποία συζητούμε, η τράπεζα NLB, είναι η μεγαλύτερη ε, σλοβανική τράπεζα που είναι ακόμα στη διεκτησία του κράτους σε δημόσια χέρια. Με φορολογικές λοιπόν ε, πλήρωμες έγινε η επανακεφαλαιοποίησή της. Την τελευταία φορά μάλιστα με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον όρο να απολυθεί στη συνέχεια η τράπεζα. Αυτή η υπόθεση λοιπόν του ξεπλήματος χρήματος, τα θέματα χορήγησης πιστώσεων σε μεγάλους παράγοντες ε, της σλοβενικής οικονομίας. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν μπορεί να αποφασίσει ο Υπουργός Οικονομικών τι θα γίνει με την τράπεζα αυτή αλλά μόνο αυτοί που είναι αναμειγμένοι στις τράπεζες αυτές εδώ και χρόνια. Πρόκειται για μια ανεξάντλητη πηγή χρήματος και πολιτικής εξουσίας στην Σλοβενία η τράπεζα αυτή. Και η ιστορία αυτή δεν είναι δυνατόν πλέον να ε, συνεχίζεται. Έχουμε τεκμήρια, έχουμε έγγραφα και το Σλοβενικό κράτο δικαίου διακυβεύεται στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε δει ότι ω τώρα οι δράσει, οι θεσμικοί, τα θεσμικά όργανα δεν έχουν καταφέρει να αντιδράσουν. Είναι σε ομοιρία, καθεστώ ομοιρία πραγματικά η σλοβενική θεσμή, όπω και ε, η Νόβα Λουμπλιάνα Μπάνκ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευρεντική επιτροπή του Σλοβενικού Κοινοβουλίου, υπό την ηγεσία του κυρίου Λόγκαρ. Χάρη στις εργασίες της Επιτροπής αυτής ξέρουμε τα ονόματα των επαιτίων πλέον και πολλοί από αυτούς είναι σε υψηλέ πολιτικές θέσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες. Άλλοι ευημερούν στην επιχειρηματική ζωή και της Σλοβενία, αλλά και στην Ελλοδαπή. και μετά ρωτάμε τον κόσμο γιατί τα πηγαίνει άσχημα, γιατί έχει τόσο χαμηλούς μισθούς. Μα μία από τις απαντήσεις είναι η NLB, η τράπεζα NLB. Η επίλυση λοιπόν του προβλήματος αυτού είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία και για το μέλλον της Σλοβενίας. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο, αγαπητέ Άντζε. Σε ευχαριστώ πολύ που έκανες αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή. Μία μικρή ερώτηση τώρα. Θα μπορούσες να μας δώσεις ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κύριε Μεκίνα, είναι ενδιαφέρον το ότι έρχεστε από μια εφημερίδα η οποία έχει διαπλοκίσει ότι φορά την ιδιοκτησία της με φορολογικούς παραδείσους. Πιστεύετε πιστεύετε στην ε, Ερευνητική Επιτροπή και στα συμπεριβληματά τη. Γνωρίζετε ως δημοσιογράφος το τι συνέβαινε και τι κάνατε σε περίπτωση που γνωρίζετε. Και μία είναι η ανησυχία μου, η μεγάλη ανησυχία μου. Ένα δισεξεπλήμενο χρήμα. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα, μία από τι μεγαλύτερε υποθέσει ξεπλήματο χρήματο στην Σλοβενία. Αν δεν ισχύει αυτό και αν δεν πρόκειται για ξεπλήμα χρήματο, γιατί πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ, ο επόμενο ομιλητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κάποια παραδείγματα ανέφερα στην παρουσίασή μου, αλλά η παρουσίαση την ε, έχετε και στα εγγραφά σας. Να σας περιγράψω όμως μία υπόθεση, επιτρέψτε μου, μία πρεσβεία. ενός κράτους της ε, Ευρώπης έκανε 500 ε, αναλήψεις χρημάτων τις οποίες και μεταβιβάστηκε σε λογαριασμούς από το 99, γιατί στη συνέχεια δημιουργήθηκαν συστήματα εσωτερικού ελέγχου στην τράπεζα και οι αναλήψεις πάνω από 1000 ευρώ πλέον καταγράφονται. Αυτά τα χρηματικά ποσά λοιπόν ε, μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό της γυναίκας του και σε τρεις δόσεις μεταφέρθηκαν τα χρήματα αυτά στην εταιρεία Φάροκο και συνεχίστηκαν ε, οι μεταβιβάσεις για διάφορα στοιχεία. Και στη συνέχεια, σε μια ευρωπαϊκή χώρα έχουμε μια άλλη ποινική δίωξη για μεταφορά χρημάτων. Ενός 22χρονου. Μια Ελλαδαπή τράπεζα εφιστεί την προσοχή στο γεγονός αυτό και παγώνει τι ε, συναλλαγέ τι μεταβάσεις αυτές. Ο άνθρωπο αυτός λοιπόν, ο, νερός αυτός πηγαίνει και σε άλλη και σε άλλη τράπεζα και σε ένα έτος έχει καταφέρει να σηκώσει ένα εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά. Αυτό που μας τρομάζει είναι ότι η τράπεζα από την οποία προήλθε μετά από τρεις-τέσσερις συναλλαγές ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία. Αλλά ο όμιλος NLB μετά από χίλιες συναλλαγές δεν προέβησε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Αυτό πραγματικά με τρομάζει. Και αυτό φοβάμαι ειλικρινά ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, κατανοήσαμε και καταλάβαμε πού ήταν το πρόβλημα. Ο κύριος Μεκίνα, και σε εσάς απευθύνθηκε ερώτηση. Like each other. Όλοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει και πάρα πολύ συμπάθεια μεταξύ μας. Δεν γίνονται έρευνες μόνο στο Κοινοβούλιο για την τράπεζα αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Στη δική μου επιχείρηση τύπου οι δημοσιογράφοι υφίστανται πιέσεις, προσπαθούν να διερευνήσουν και τις δικές μας ενέργειες. Θα ενημερώσουμε φυσικά για την υπόθεση αυτή την Διεθνή Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων. Κύριε Σλόγκαρ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσω. Η δική μου ερευνητική επιτροπή δεν έρευνα ε, τα μέσα ενημέρωση. Ούτε υπάρχει κάποια οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον κύριο Μακίνε. Πρώτη φορά τον βλέπω στη ζωή μου. Η Ερευνητική Επιτροπή έχει ω καθήκον πραγματικά να ερευνήσει τέτοιε υποθέσει. Και η υποψία για... και η κατηγορία για ξέπλυμα χρήματο αποτελεί ένα σωστό λόγο έρευνα. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι γεγονός και σημαντικό μάλιστα γεγονός ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου. Κάνετε και άλλες έρευνες, ε, τις οποίες και ακολουθείτε προφανώς εξίσου ε, έντονα. Κύριε Μακίνα. Κύριε Μακίνα. Είπατε ότι το θέμα αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό από αντίστοιχες περιπτώσεις. Ποιες είναι οι περιπτώσεις αυτές οι τόσο σημαντικές. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ε, διαφημίζουν την υποδοχή νέων επιχειρήσεων στη Σλοβενία. Ποιοι είναι οι λόγοι που γίνεται κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καταρχάς, την ερώτηση ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα ε, με τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτή ή μια άλλη υπόθεση ή κάποια άλλη υπόθεση. Εδώ και αρκετά χρόνια η Σλοβενία ήταν σε μια δύσκολη οικονομική θέση. είχε περάσει σε διαδικασίες ιδιωτικοποίησης κάποιων επιχειρήσεων διαχείρισης υποδομών. Το ανησυχητικό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι είχαν αλλάξει οι νομικές ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μπορούν να απολυθούν και σε α, επιχειρήσεις offshore. Μέχρι τότε οι κυβερνήσεις μπορούσαν να πουλήσουν σε επιχειρήσεις των οποίων ήταν ξεκάθαρα το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αλλά όταν ήρθε αυτό το νέο κύμα ιδιωτικοποιήσεων μπορούσαν ε, ε, υποδομές να πολιθούν και σε εταιρείες με έδρα τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό που αρκούσε ήταν να κάνουν μια δήλωση οι ε, αγοραστές ότι είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Οι εξηγήσει τις οποίες έδωσαν τα κυβερνητικά όργανα ήταν ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, μπορούν οι κρατικές επιχειρήσεις να πολιθούν ε, με υψηλότερο τίμημα σε εταιρείε από φορολογικού παραδείσους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με τα τεστ κοπόσεως των σλοβενικών τραπεζών, με τις κόκκινες εισαγωγικά τράπεζες, αλλά ακόμα και οι εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν τα stress test της τράπεζες είχαν έδρα τους φορολογικούς παραδείσους. Νομίζω ότι το σύστημα offshore ε, τελικά δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση κάθε φορά όπως η NLB. Είναι κάτι το οποίο είναι αν θέλετε η ψυχή και ο πυρήνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο κύριος Λογκάρ. Ευχαριστώ και φυσικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση. Όταν μιλάμε για τέτοια υποψία του δρόμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο πρωθυπουργός, ο Υπουργό άμυνας, ο Υπουργό ε, Εσωτερικών, ο Υπουργό Οικονομικών, όλοι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί με έκθεση του δυσιογραφικού πρακτορείου. Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει οργανωθεί μια συνεδρίαση. Τίποτε όμως δεν συνέβη. Η ηγεσία του κράτους ήταν ενημερωμένη. Τίποτα δεν διοργανώθηκε όμως. Δεν έγινε καν συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Ερευνητική Επιτροπή, ε, εξετάσαμε τα θέματα αυτά και περιλαμβάνονται και τα πιο σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια τεράστια υπόθεση. Αλλά και πάλι τα πορίσματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό. Η Διερευνητική λοιπόν Επιτροπή αποτελεί μια απόπειρα διορθωτική αν θέλετε. Να διορθωθεί κάτι. Και διαπιστώσαμε ότι ο μηχανισμός ε, εποπτεία, στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργήσε στη Σλοβενία. Αυτό που ελπίζουμε τελικά είναι πλέον να είμαστε βέβαιοι για τα γεγονότα και να βελτιώσουμε, να έχει βελτιωθεί πλέον το σύστημα, προκειμένου να μην παρασιάζονται τέτοια φαινόμενα πλέον. Ο κύριος Λογκάρ είπε ότι όλοι οι σημαντικοί πολιτικοί στην Σλοβενία γνώριζαν για την υπόθεση αυτή. Εγώ πριν προσπάθησα να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την υπεύθυνη υπάλληλο να αντιμετωπίσει συνολικά και να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά αν όλοι οι πολιτικοί γνώριζαν για τα θέματα αυτά, να θέσω και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν από το κόμμα του κ. Λόγκα. Ο υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών είχε διοριστεί από το κόμμα του κυρίου Λόγκαρ. Ο υπεύθυνο για την διαχείριση της NLB, ε, ο υπεύθυνο εννοώ για τις ε, συναλλαγές αυτού του τύπου, είχε επίσης διοριστεί από την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε το κόμμα του Λόγκαρ. Και ήδη από το 2012 όταν άρχισαν οι Γάλλοι να κάνουν ορισμένες έρευνες για την NLB, έστειλαν επιστολές ε, ε, στο Υπουργείο, στον Υπουργό, ο οποίος ανήκε ε, φυσικά στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε το κόμμα του κυρίου Λόγκαρ. Το ερώτημα του ποιο δεν ανέλαβε τι ευθύνε του και τα κοντά του δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εδώ. Εμεί θέλουμε αυτή τη στιγμή να εγκαθιδρύσουμε να δούμε ποια είναι τα, περιθετικά. περιστατικά. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πιο πολλές πτυχές από ό,τι φαινόντουσαν ε, εκ πρώτης όψεως και ενδεχομένω να πρόκειται και για συστημική, ε, συστημικό παράπτωμα και αμέλεια. Κύριε Λόγκαρ. Κοιτάξτε, υπήρξαν άμεσες κατηγορίες τις οποίες οφείλω να ανατρέψω. Όπως είπαμε, η εισαγγελία δεν ήταν ενημερή. Όταν η εισαγγελία δεν είναι ενήμερη, δεν μπορεί να δράσει. Είναι ανεξάρτητη η εισαγγελία στην Σλοβενία. Ούτε ο υπεύθυνο των μυστικών υπηρεσιών ήταν ενήμερο. Η δε κυβέρνηση του α, Πρωθυπουργού ενημερώθηκε. Η κυρία Σκοτ Κάτω για του πράσινου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα συνεχίσω μετά την ερώτησή σας, Πρόεδρε, λέει η κυρία Κέιτο. Υπήρξαν και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες ότι υπήρξαν παραβιάσεις από πλευράς της NLB ε, των υποχρεώσεων της να ε, ε, ανοιχνεύσει την έδρα των δικαιούχων των λογαριασμών που προχώρησαν στο πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Σαν παράδειγμα δεν προχώρησε στον έλεγχο της πηγής του πλούτου του κυρίου Φαροξαντέ, του βασικού καταθέτη. Δυστυχώς σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ε, πλησίματος βρώμικου χρήματος δραστηριοποιούνται και διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο City του Λονδίνου. Ε, κάποια από τα χρήματα αυτά μήπως πήγαν στο City, μήπως πήγαν σε ιδιοκτησίες στο Λονδίνο, μήπως πήγαν σε ρωσικές τράπεζες στην Αγγλία. Ο κύριος Μακίνα. Πράγματι τα χρήματα πήγαν σε πάρα πολλές μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ακριβώς το τι είχε συμβεί και οι πιο λογικές εξηγήσει είναι ότι επειδή οι μεγάλες τράπεζες είχαν τιμωρηθεί από τη ΣΥΠΑ και επειδή οι ΙΠΑ το 8 άλλαξαν την ερμηνεία των νομικών ρυθμίσεων και ξεκίνησαν επιβολές κυρώσεων εξωτοπικές των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλοί Ιρανοί πήγανε σε μικρές τράπεζες και μέσω των μικρών τραπεζών έστελαν τις καταθέσεις τους στις ε, μεγαλύτερες ευρωπαϊκές. Μια άλλη δήλωση. Αυτά τα οποία λέω εδώ αναφέρονται στις γενικές τάσεις. Εγώ δεν λέω ότι κάθε μία από τις συναλλαγές αυτές ήταν ξεκάθαρη. Πολλές από τις συναλλαγές κρύβουν πάρα πολλές επιχειρήσεις κρύβουν πάρα πολλούς δικαιούχους και έχουμε κάποια παραδείγματα. Ξέρω ότι η Γαλλία ελέγχει μια περίπτωση τραπεζικής απάτης στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Λόγκαρ. Αλλά αν θέλουμε να κατανοήσουμε γενικά το τι συμβαίνει, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο με τη λογική αυτή και η συζήτηση μπορεί περισσότερο να γίνει ανάμεσα στα κράτη και στο Ιράν. Έχετε και άλλη ερώτηση, συνάδελφε. Okay, please. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πιο πολλά από αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην ε, Γερμανία και η Ιταλία αναφέρεται και η Μεγάλη Βρετανία η Γαλλία αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι τα άτομα τα οποία έλαβαν τα χρήματα αυτά στη συνέχεια διώχθησαν από τις εκάστοτε χώρες λόγω ζητημάτων ασφάλειας ή λόγω ποινικών διώξεων. μετά από αποπίεσει ε, αναστάλησαν οι δικασίε αυτές και μεταφέρθηκαν πολλά χρήματα και σε ρωσικούς ομίλους. Και σε επανειλημμένες περιπτώσεις οι τράπεζες αρνήθηκαν να συνεχίσουν τις συναλλαγές, γιατί πραγματικά είχαν δυσκολευτεί, είχαν δυσκολέψει αυτές οι συναλλαγές. Τι γίνεται όμως με την απώλεια και την αποτυχία της δέουσας επιμέλειας και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Προφανώς υπάρχουν σαφείς ε, ε, διατάξεις, ε, ελέγχθη σε ποια δράση. Είναι τεχνική ερώτηση. <clears throat> Είναι πολύ δύσκολο. Η ερμηνεία της Ευρώπης τότε ήταν εφόσον δεν επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν οι κυρώσεις ε, δύο ευρωπαϊκών τραπεζών ε, σε συνονίσεις μεταξύ τους προς το Ιράν μπορεί να ήταν ε, εντάξει αλλά όχι από την Ευρώπη συνολικά προς το Ιράν διότι δεν επέβαλε κυρώσεις η Ευρώπη στο Ιράν αλλά η ΕΠΑ. Κάποια στιγμή η ερμηνεία άλλαξε, οι νόμοι άλλαξαν και υπόθηκε ότι ακόμη και αν το Ιράν κάνει συναλλαγές με το Βερολίνο και το Παρίσι σε δολάρια, αυτό μπορεί να αποτελεί παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ήταν ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, πολύ περίπλοκες διατάξεις, όπως θα έχετε δει και πριν από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Προφανώς είναι πολλοί δικηγόροι, νομικοί χώρες που τα σκέφτηκαν αυτά και κοιτάζουν πώς θα ορίσουν το τι είναι νομιμοποίηση παράνομα προσόδων, τι δεν είναι και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ και τώρα έχουμε ακόμα τρεις ομιλητές στον κατάλογο. Ο πρώτος. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα να βγάλω από όλα αυτά. Μου φαίνεται πραγματικά σαν καταγίδα κρανίο. Βεβαίως η αμερικανική πολιτική για το Ιράν είναι γνωστή αλλά μου φαίνεται ένα πρόβλημα ε, αστυνομία και δικαστών στη Σλοβενία. Γιατί δεν αντιδράσανε, γιατί δεν τα καθαρίσανε οι ίδιοι οι Σλοβαίνοι. Δεν θα έπρεπε η ίδια η Σλοβένικη κυβέρνηση να τα ερευνήσει. Τι σχέση έχει αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαφέρον είναι που έχουμε οργανώσει ακρόαση, αλλά θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα κράτου μέλου αυτό, του ίδιου του κράτου μέλου, όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που χώνεται με τη παντού στι δουλειέ των αλωνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει κάτι να βρει να έχει να κάνει και παρεμβαίνει στα πάντα για να δικαιολογήσει την τεράστια γραφοκρατία της και τους παχυλούς μισθούς των ανθρώπων σε αυτό το κτίριο. Θα πρέπει κάπως να αντισταθούμε στην ε, παρεμβατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τράπεζες να ε, συνεχίσουν να λειτουργούν ε, άνετα αλλά χωρίς τον καπιταλισμό που βασίζεται σε σχέσεις προτιμησιακές. Πολλά ε, ποσά ε, πέρασαν και από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά είναι μεγάλο ε, μέρος της ευαισθητότητάς μας αυτό. Είναι πολλά τα ποσά που πήρατε από εμά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει και άλλα από το Βρετανό φορολογούμενο. Διαρκώ κατηγορείται το City του Λονδίνου. Ως Βρετανός πολίτης και Βρετανός εκπρόσωπος του λαού μου το βρίσκω επωνίδιστο αυτό. Αλλά πραγματικά δεν πολύ καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Εδώ νομίζω ότι απλώς κατασπαταλούμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ντέβιντ έδωσε έγκριση για τον κύριο Κλήρινγκ στην ε, Ευρώπη και όχι στο Λονδίνο. Ποιος έχει απάντηση στην ερώτηση αυτή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να υποδείξω το εξή στην περίπτωση Τη αποτροπή ε, ξεπλήματο βρωμικού χρήματο. Δύο πράγματα θα πρέπει να εξετάσουμε σε ό,τι αφορά την υποψία ε, για υποθέσει ξεπλήματο χρήματο και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και γι' αυτό λοιπόν ανέφερα μία περίπτωση στην εισαγωγή μου. Έχουμε 2.000 ε, πελάτες, μάλλον 2.000 λογαριασμούς ιδιωτών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 100 δις ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω και το εξή. Μας προσκαλέσατε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ, σας είμαι ευγνώμων. Αν ε, τα θεσμικά όργανα της Σλοβενία ε, είχαν αντιμετωπίσει με τον δέοντα τρόπο την υπόθεση αυτή, δεν θα είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, θα είχαμε βρει μια λύση. και ένα μέλος της Επιτροπής Καταπολέμησης της ε, Διαφθοράς πριν ολοκληρώσει την έρευνά του έλαβε θέση στην ε, NLB και ασχολείται με θέματα συμμόρφωσης πλέον στην τράπεζα NLB. Δουλειά του δηλαδή είναι να διαπιστώνει πώς οι πληροφορίες για το ξάπλυμα βρώμικου χρήματος ε, κατέληξαν τελικά στη, δημόσια, στη δημοσιότητα. Τα άτομα τα οποία που έλαβαν τις πληροφορίες από τη μυστική υπηρεσία είναι πλέον πρωθυπουργός. Ο κ. Βόγκα, ο οποίος ήταν υπουργό εξωτερικών, είναι ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ευρωπιτροπής στο Κοσφοπέδιο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Διαφθοράς, ο οποίος ενημερώθηκε από πληροφοριοδότες, είναι σήμερα υπουργό δικαιοσύνη και είναι υποψήφιος της Σλοβενικής Δημοκρατίας για Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας είπα τι χρηματικά ποσά κατέληξαν στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας παρουσίασα πως τμήμα τουλάχιστον των χρημάτων αυτών είναι ύποπτης προέλευσης. Και νομίζω ότι αυτό σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Okay, just <clears throat> the, the, the police was, of course... Η αστυνομία ερευνούσε βεβαίως την όλη υπόθεση, όπως είπα προηγουμένω. Και βάσει των πηγών μα ήταν σε επαφή με όλη τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή τους φορείς που ασχολούνται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Απλώς δεν μπορούσαν μόνοι τους να λύσουν το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής μόνοι τους. Σας ευχαριστώ. Δύο άτομα ζητούν το λόγο. Θα ήθελα να πω κλείνοντας το εξή. Πρόεδρε, εδώ λοιπόν το clearing θα έπρεπε να γίνεται στην Ευρώπη και όχι στο Λονδίνο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε βγάλει άκρη. Διότι δεν θέλουμε αυτόν τον παρεμβατισμό από μια χούφτα γραφειοκράτε τη Βρυξέλλε που καταστρέφουν ε, το εμπόριο. Δεν θέλουμε να γίνουμε κάλαθο αχρήστων ε, για όλε τι συναλλαγέ τη υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι άλλη ημέρα το θέμα. Ο κύριο Χέι από το ΕΛΚ και μετά ο Μίλαν Σβέρο, τελευταίο ομιλητή για το γύρο των ερωτήσεων αυτών. Brian και να διευκρινίσω ότι έχουμε πέντε λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Και σε κάτι που έθεσε η αντιπρόεδρο η κυρία Γκόμες προ τον κύριο Μεντίνα. Έκανε λόγο προηγουμένω για άλλε υποθέσει. Εξίσου σοβαρέ ή και σοβαρότερε από αυτήν. Από το να μας λέτε παρουσία σα για τι πωλήσει των ε, περιουσιακών στοιχείων και πώ πήγαν αυτά offshore. Μπορείτε να δώσετε τρει συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των σοβαρών υποθέσεων. Αυτό θα μα ενδιαφέρε. Δεύτερον, για το θέμα τη Ερευνητική Επιτροπή. Ε, σα ασκήθηκε πίεση και στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή τη στιγμή της έρευνας για το πώς θα κάνετε τη δουλειά σας και μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το από πού προήλθε αυτή η πίεση από διάφορε πλευρέ, φαντάζομαι, του σλοβενικού κράτου. Και μια τελευταία ερώτηση. Με το παράδειγμα των γαλλικών αρχών που ασχολήθηκαν μια περίοδο, περίπτωση απάτη, όπου υπήρχαν πολλαπλοί λογαριασμοί σε πολλαπλέ τράπεζε. Ήταν αυτή η μόνη υπόθεση που έχετε εντοπίσει ω τώρα, διότι οι γαλλικέ αρχέ, η μόνη αρχή που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό ω επίπτωση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο, έχει αναλάβει διαφορετική δράση. Ευχαριστούμε κύριε Μεντίνα, εσεί πρώτο. Ναι, πολύ συγκεκριμένα. Με το κύμα ιδιωτικοποιήσεων στη Σλοβενία σχεδόν κάθε, κάθε πώληση περιουσιακού στοιχείου φύγανε σε offshore, όπως το Λουξεμβούργο, έτσι, ενώ και αυτές τις περιπτώσεις. Η δεύτερη τραπεζά μας πουλήθηκε σε Λουξεμβούργιο, σε Λουξεμβούργιο. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι διοκτήτες. Άρα το κράτος ευχαριστιέται αν πάρει κάποια ενυπόγραφη δήλωση ότι είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες. Δεν κοιτάνε που είναι καταγεγραμμένοι αυτοί. Δεν χρειάζεται πλέον κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά να είμαστε σαφείς, διότι χρησιμοποιήσατε το επιχείρημα μόλι σας, μόνο σας, ε, ταξινόμηση κάνατε. Ε, πείτε μας τρία παραδείγματα Πείτε μου τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις, αντί να μου λέτε διάφορες εξηγήσεις. Μόλις σας το είπα. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζά μας. Τα περιουσιακά στοιχεία τώρα δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις εταιρείες. Της DGC. Ε, Σλοβενικής εταιρείας με που πουλήθηκε σε Αμερικανούς. Τι είναι αυτές οι υποθέσεις ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Δεν μιλάω για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάω για παρατήρηση. Για φοροαποφυγή. Βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι φοροαποφυγή αυτό αν είναι Λουξεμβούργο. Ο κύριος Σφέαρ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ τον ε, Δόκτωρ Λόγκαρ για την εργασία του και για τις αφέστατε απαντήσει του. Θα είχα μία ερώτηση ακόμα να κάνω. Από το 2014 στην Ευρώπη υπάρχει ένα μηχανισμό ε, ένας μηχανισμός για την προστασία του κρατου δικαίου. Ε, ο οργανισμός αυτός ε, προβαίνει σε συστάσεις, ε, σε μέτρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγύηση για το κράτος δικαίου σε κάποια χώρα. Η ερώτησή μου είναι, είναι σε θέση η Σλοβενία να λύσει το θέμα αυτό ή όχι, ή θα χρειαζόταν παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Και κοιτάξτε, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημα κατά να ασκήθηκε πίεση ή όχι. Εγώ είμαι διπλωμάτης και έχω διπλωματικό καθεστώς. Δεν ξέρω κατά πόσον υπήρξε πίεση υπό την έννοια αυτή ή όχι. Απελγηθήκαν μέχρι και οι γονείς μου. Η Ερευνητική Επιτροπή συχνά χάνεται στα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, μετά την ανακοίνωση τύπου για την έκθεση της Επιτροπής μας. Επί δύο ημέρες ε, δημόσια, στα δημόσια μέσα ενημέρωση δεν αναφέρθηκε τίποτε σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Η Επιτροπή μας διαπίστωσε πάρα πολλές ε, ελλείψεις, πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είμαι εγώ σε θέση να κρίνω κατά πόσο η Σλοβενία και θεσμική, ε, τα θεσμικά της όργανα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε τέτοιε περιπτώσεις. Ελπίζουν να είναι σε θέση. Υπάρχουν κάποιοι σχετικοί δείκτες, αλλά προφανώς ε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να ερευνήσουν τις περιπτώσεις αυτές, τις υποθέσεις αυτές, τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στις έρευνε του 2010 και δεν κατέληξαν σε οποιοδήποτε συμπέρασμα θα πρέπει φυσικά να αντικατασταθούν από άλλους υπεύθυνου. Δεν ισχύει. Δεν έκαναν σωστή και ανταλλαγή έρευνα των υποθέσεων αυτών. Και μιλήσαμε και με πολλούς από τους ερευνόμενους και μας επιβεβαίωσαν ότι δεν επικοινωνούσαν καν μαζί τους η αστυνομία. Επειδή είσαστε μέλη της Εθνοσυνέλευσης, το διπλωματικό καθεστώς αναγνωρίζεται αυτόματα. Το σε trenutkom, ko smo začeli zaslišati priče pred preiskovalni komisiji. Κοιτάξτε, mi στιγμή που κάναμε kresto na martiron. και αποκαλύφθηκε ότι τα προσόντα του καθενό ήταν πιο υψηλά από ό,τι χρειαζόταν για την ε, εκάστοτε θέση. Εγώ να σα πω ότι μιλάω για δύο υποθέσει. Μία είναι ήδη επιτυχηση ή η άλλη δεν έχει ακόμα καταλήξει σε συμπέρασμα. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να πάρω το λόγο. Μάλιστα, πολύ ωραία και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω στην περίπτωση αυτή, λέει ο πρόεδρο. Δεν τα διευκρινίσαμε όλα, αλλά κατανοήσαμε ότι υπήρξαν ε, μηχανισμοί οι οποίοι οι οποίοι προώθησαν το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος ε, και ήταν τρομοκρατικές ε, ενέργειες αυτές οι οποίες ε, χρηματοποτήθηκαν και τελικά αποκάλυψαν την υπόθεση αυτή. Τα γαλλικά αιτήματα, οι έρευνε του Σλοβανικού Κοινοβουλίου δεν το διευκρινίσαμε αυτό και σε ό,τι ισχύει και για την αμερικανική πλευρά θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Λεγκόρη, κύριε Μεκίνα, τους συναδέλφους, τα εκκρεμία αυτά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να λάβουν απαντήσεις ε, και στην Σλοβενία. Τέτοια πολιτικά ζητήματα δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εδώ πέρα, ούτε όπως την υπόθεση του Λουξεμβούργου, της Μάλτας. Πρόκειται για πολιτικά τέτοια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα διελευκάνουν οι ίδιες οι χώρε. Σα ευχαριστώ και θα κλείσω το πάνελ αυτό στην προηγουμένη περίπτωση. Να κάνουμε ένα διάλειμμα 4 λεπτών. Και έχουμε ήδη του ομιλητές του επόμενου πάνελ μαζί μα Να κάνουμε μια, ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε 4 λεπτά. Bitte Platz nehmen. Ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε με μια ελαφριά καθυστέρηση το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο πάνελ Αζερμπαϊτζάν σε ό,τι αφορά τις ε, αποκαλύψεις λάτμα και θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας. Πρώτος ε, ε, είναι ο Καλντόλαν, ο οποίος είναι της, ο Καλντόλαν, διευθυντής της Transparency International στις Βρυξέλλες και δύο δημοσιογράφοι από την δανική εφημερίδα Berlingske, Εύα Μίχαλ Λούντ Τρει συγγνώμη, δημοσιογράφη και ο Σάιμον Μπέντσεν τρίτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήλθατε εδώ σήμερα και είδατε ζωντανά πώς ε, θα εκτελεχθεί η συζήτηση, θα έχουμε καταρχά τι ε, παρουσιάσει, καταρχά από του δημοσιογράφου. Ποιο θα πάρει το λόγο, ο κύριο Λούντα από μέρου σα. Θα ξεκινήσετε και μετά το λόγο έχει ο κύριο Ντόλαν. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία από το λεγόμενο Λάντροματ, το πλυντήριο του Αζερβαϊτζάν. Η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες ε, υπηρεσίες τύπου ξεκίνησε μετά από παρατηρήσεις διακίνησης χρημάτων ανάμεσα σε ε, δανέζικες τράπεζες, κυρίως την Danske Bank, μια από τις μεγαλύτερες, και εσθονικές τράπεζες. Υπήρχαν προβλήματα στις τράπεζες αυτές σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στον κανονισμό AML, ιδιαίτερα γύρω από τις συναλλαγές που μπορεί να έχουν σχέση με πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Οι πελάτες όταν κάνουν ύποπτες συναλλαγές κρύβονται πίσω από offshore επιχειρήσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε αυτή η απόκρυψη αν θέλετε και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι τις παράνομες δραστηριότητες. Είδαμε πως το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν πέρασε εκατομμύρια από ε, την τράπεζα Ντάνσκε ε, για να δωροδοκίσει τοπικούς πολιτικούς, για να επηρεάσει ευρωπαίους πολιτικούς και για δώρα και εξαγορές. Similar cases of suspicious activities such as money laundering and tax evasions, the masterminds used British LP or LLP companies in this... Χρησιμοποιήθηκαν κάποιες ε, επιχειρήσεις γέφυρα θα έλεγα για να κυκλοφορούν τα χρήματα αυτά. και για να φέρουν εις πέρας ακριβώς ε, τις παράνομες δραστηριότητές τους. Είναι θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση στη Δανία. Ε, δεν μπορούσαμε να βρούμε φυσικά εύκολα τα ονόματα των δικαιούχων των λογαριασμών. Βλέπετε κάποια επιμέρους στοιχεία. οι επιχειρήσεις που έλεγχαν τις επιχειρήσεις που είχαν τους λογαριασμούς στην Τάνσκε είχαν έδρα σε διάφορες περιοχές του κόσμου όπως τις Βρετανικές Παρθένες νήσους. Υπήρξαν τέσσερις επιχειρήσεις ε, οι οποίες είχαν εμπλακεί και σε ε, προσπάθειες δωροδοκίας πολιτικών και στην Ιταλία και σε δώρα προς πολιτικούς στα πλαίσια της εκλογής του αντιπροσώπου του Αζερμπαϊτζάν σε θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι τέσσερις επιχειρήσεις λοιπόν μετέφεραν σε μια Ιταλική επιχείρηση η οποία ελέγχεται από τον Λούκα Βολοντέ τεράστια ποσά. That these four companies in fact worked as so-called slush funds ήταν τα λεγόμενα slash funds, τα οποία ελέγχονται από το καθεστώς του Αζερβαϊτζάν. Και αυτό μας έκανε να ελέγξουμε τις 16.000 συναλλαγές και να δούμε τους δικαιούχους. Ο συνάδελφος εδώ θα σας δείξει κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Η προέλευση των εκατομμυρίων που πήγαν στην Εσθονική τράπεζα της Ντάνσκε όμως ε, ήταν δύσκολο να βρει κανείς, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει σωστά τους δικαιούχους, είδαμε όμως ότι είχαν κάποια σχέση με το Αζερβαϊτζάν. Αναλύσαμε τους τέσσερις λογαριασμούς των τεσσάρων αυτών εταιριών και είδαμε ότι πάρα πολλά χρήματα προήλθαν απευθείας από το καθεστώς του Αζερβαϊτζάν. Ας πούμε από την ε, ε, Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων και επίσης ε, την Υπηρεσία Προστασίας που συνδέεται άμεσα με τον πρόεδρο Αλιεφ επίσης και από κάποιες μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις ή ισχυρούς αζέρους οι οποίοι έχουν στενές σχέσεις με το καθεστώς. 1,4 δις από την Μπακτέλεκομ η οποία από ό,τι φαίνεται ταυτίζεται ε, με μια εταιρεία Telecom αλλά στην ουσία δεν έχει κανένα περιεχόμενο και δημιουργήθηκε από τον Άζαντοφ, τον γιο του προηγούμενου ε, Υπουργού Ενέργειας. Υπήρχαν βέβαια και άλλες επιχειρήσεις που είχαν συμβάσεις με το κράτος του Αζερβαϊτζάν. Πολλές από τις ε, συναλλαγές αυτές προήλθαν και από την Κεντρική Τράπεζα ε, του Αζερβαϊτζάν που ελέγχεται φυσικά από την κυβέρνηση. 29 εκατομμύρια προήλθαν από την Ρωσομπόρ, η οποία είναι ε, κρατική ρωσική εταιρεία που εμπορεύεται όπλα και στην ουσία ήταν μετά από αγορές που έκανε το Αζερβαϊτζάν μίζες προς υπεύθυνους αζέρους αξιωματούχους. Ε, η έρευνά μας χαρακτηρίστηκε προκλητική και αστήρικτη από το καθεστώς. Τώρα θα σας παρουσιάσει ο συνάδελφος κάποιους από αυτούς που ωφελήθηκαν από αυτές τις ε, ενέργειες. Αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί μέσω του Λόντροματ, όπως ονομάστηκε το Αζερβαϊτζάν, έλαβαν χρήματα. Από το 2016 που να αναλύουμε τα ποσά, βρήκαμε πολλά χρήματα να ε, μεταφέρονται με τα τσουβάλια σε αυτούς τους πολιτικούς κάποιες φορές. Τους ε, ερευνήσαμε αυτούς τους ε, πολιτικούς και υπαλλήλους που είναι ψηλοί αξιωματούχοι και είχαν κάτι κοινό. Ε, ότι μιλούσαν με τον ίδιο τρόπο για αυτού του είδους το σύστημα, ενώ το Αζερβαϊτζάν θεωρείται ως ένας, ε, μια από τις χώρες που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μπορούσε να θεωρηθεί και δικτατορία, οι πολιτικοί αυτοί μιλούσαν υπέρ του καθεστώτος. Να αναφέρω μερικούς από αυτούς τους ισχυρούς. Έντουαρτ Λίτνερ, ε, πρώην μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και πολιτικός πολλά χρόνια, ο οποίος υπερασπίστηκε το Αζερβαϊτζάν ε, επίσης ε, στον ΟΑΣΕ ε, που οι εκλογές του 2013 θεωρήθηκαν ανελεύθερες και μη δημοκρατικές, ο κύριος Λίντνερ τις, υπος, τις παρομοίασε με τις δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές στη χώρα του, στη Γερμανία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο κύριος Κάλιν που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και ήταν παντρεμένος με την ε, πρόεδρο της UNESCO μέχρι πρόσφατα. Το ζευγάρι αυτό ε, μέσω της UNESCO ας πούμε απένει με χρυσό μετάλλιο στον ε, αντιπρόεδρο της χώρας που ήταν πρωθυπουργός και έχει επενέσει το Αζερβαϊτζάν που προέ προήγε την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου ε, στο επίπεδο της UNESCO. Ενώ ξέρουμε ότι οι επιδόσεις του Αζερμπαϊτζάν σχετικά είναι πολύ χαμηλές. Είναι πολλοί οι πολιτικοί που έχουν λάβει χρήματα από αυτό το σύστημα ε, και όλοι αρνούνται ότι δωροδοκήθηκαν αλλά δεν έχουν καμία λογική εξήγηση για το λόγο ε, που αυτές οι συναλλαγές έγιναν με τρόπο μυστικό και κρυφό. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι πολλοί υψηλοί αξιωματούχοι του Αζερβαϊτζάν ανά τον κόσμο έλαβαν χρήματα ή φρόντισαν να στείλουν χρήματα σε όσους ε, είχαν άμεση σχέση με το Αζερβαϊτζάν, έστω και μέσω της οικογένειάς τους. Για τις συναλλαγές αυτές που ερευνήσαμε, ε, βρήκαμε πολλούς από τους δικαιούχους, αλλά και κάποιους άλλους, ε, κάποιοι άλλοι παραμένουν ανώνυμοι. Και Υπάρχει υλικό το οποίο δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε ακόμη σήμερα. Επίσης για τις πιθανές διασυνδέσεις με τη Μάλτα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μάλτας έχουν αναφέρει ένα πρόγραμμα λεύκανσης προσόδων όπου εταιρείες από, μάλλον τράπεζες από το Αζερβαϊτζάν αγοράζουν εταιρείε αυτοκινήτων λόγου χάρη που έχουν σχέση με πολιτικούς ε, κάποιες φορές. Δεν έχουμε βρει στο υλικό μας όνοματα εταιρεών και τραπεζών, αλλά οι διαδικασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί μοιάζουν. Πολύ σύντομα λοιπόν για τη συνέπειες ανά την Ευρώπη βλέπετε τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Κάποιοι πολιτικοί ζήτησαν έρευνες, έχουν ξεκινήσει δηλαδή σχετικές έρευνες σε πολλά ε, μέρη της Ευρώπης και τελική παρατήρηση αυτή η φωτογραφία. Φωτογραφία ενός σπιτιού ε, έξω από τον Μπακού ε, στο Αζερβαϊτζάν. Ο άνθρωπος που ζει σε αυτό το ταπεινό σπίτι είναι δικαιούχος δύο από, τον, από αυτούς τους βασικούς λογαριασμούς ο άνθρωπος που ζει σε αυτό το σπίτι θα μπορούσε να είναι επικεφαλής εταιρεία με ροές ε, πάνω του ενός δις ευρώ. Οι πελάτες, εφόσον δεν ήταν γνωστοί, θα έβλεπαν ότι ο άνθρωπος που ζει εδώ δεν είναι ούτε εκατομμυριούχος ούτε δισεκατομμυριούχος. Απλώς κρύβει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα τους πραγματικούς ενόχους και αυτούς που ωφελούνται. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Μας δώσατε πολλά παραδείγματα. Η Κάριν Στρέντς από την Ομοσπονδιακή Βουλή ε, μας έχει αποστείλει γραπτή γνωμοδότηση ε, και μας λέει ότι οι δραστηριότητες από τις 3 Ιουλίου 2014 ως σήμερα το 2017 και επειδή είναι επικεφαλής της ε, ομάδας φίλων, εκεί καταγράφεται, Και ε, εκεί έχει γίνει η όλη προσπάθεια επιρροή. Τέτοιε ομάδε φίλων έχουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο και υπάρχει σε πολλέ βουλέ. Θα πρέπει να αναλύσουμε αυτέ τι περιπτώσει πολύ προσεκτικά. Τα έγγραφα σα έχουν διανεμηθεί, να τα κοιτάξετε. Δεν έχουμε κάποια γνώμη σχετικά προ στιγμήν. Αλλά ο κύριο η κυρία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κύριε Ντόλαντ, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε λοιπόν τα θέματα μας. Είμαι ο Καλ Ντόλαν, είμαι υπεύθυνο του Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της Transparency International, η οποία ηγείται της μάχης κατά της διαφθοράς στον κόσμο. Εμείς προσπαθούμε να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τις επιπτώσεις της ε, διαφθοράς εδώ και 24 χρόνια. Έχουμε καθιερώσει τον ετήσιο δίκτυ αντίληψης διαφθοράς και το Αζερβαϊτζάν είναι ε, στις 100 χώρες η 300. είναι ένα σκορ, ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει πράγματι υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Όλα αυτά είναι γνωστά από τις διεθνείς οργανώσεις, από τους ανεξάρτητους επαγγελματίες ερευνητές δημοσιογράφους και υπάρχουν συνέπειες στους κατοίκους του Αζερβαϊτζάν όπως το θέμα της απώλειας πολιτικών ελευθεριών. Υπάρχουν όμως και επιμολύνσεις από την διαφθορά αυτή υπάρχει διαφθορά η οποία εξάγεται συστηματικά από το αζέρικο καθεστώς και στις δυτικές χώρες όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπονομεύει την ακαιρεότητα επίσης των χρηματαγορών και άλλων αγορών. Πέραν του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βασική εξαγωγή της χώρας αυτής είναι η διαφθορά. Ε, θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στις μορφές επιμόλυνσης που επηρεάζουν και τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Το πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διευκολύνει το πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Οι λεγόμενες κούφιες εταιρείε ε, είναι αυτές τις οποίες χρησιμοποιεί μεθοδολογικά Υπήρξαν τέσσερις τέτοιες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν λογαριασμού στην Εστονία 2,5 δις ευρώ, 16.000 συναλλαγές έγιναν αντικείμενο επεξεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κανένα εμπόδιο. Κανένας δεν ζήτησε πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες και τους δικαιούχους των λογαριασμών αυτών. Το οργανωμένο έγκλημα και οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι δεν χρειάζεται να δημιουργούν λογαριασμούς και επιχειρήσεις σε offshore εταιρείε, αλλά μπορούν να το κάνουν στο εσωτερικό της Ένωσης. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το λάντροματ, το αζέρικο, θα μπορούσε να συμβεί για μια ακόμη φορά στην Ένωση. Η απάντηση είναι καταφατική. Πρώτον, είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει κανείς μια τέτοια κούφια εταιρεία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε και στην Ολλανδία σε σχέση με τα Paradise Papers. Το αζέρικο λοιπόν λάντρωμα δεν είναι μια απομονωμένη περίπτωση. Οι συνάδελφοι στην Transparency International του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσαν ε, μια έκθεση λέγοντας ότι ε, ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται ε, αλλά και είναι φανεροί από όλους. Η έκθεση αυτή εντοπίζει 52 περιπτώσεις διαφθοράς που εμπλέκουν 766 αγγλικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο ελκυστικό. Μικρό κόστος εκκίνησης ε, ε, επιχειρήσεων, ταχύτητα και νομοθεσία που προσδίδει νομιμότητα, αν θέλετε, στις επιχειρήσεις αυτές κοστίζει μόνο 12 λίρες το να ιδρύσεις μια τέτοια επιχείρηση και χρειάζονται λίγα λεπτά. Ενώ κοστίζει 1020 ε, ε, ε, λίρες και χρειάζονται 90 μέρες για να δημιουργήσεις μια τέτοια επιχείρηση στις Βρετανικές Παρθένες. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν είναι η ηγέτης στο να δημιουργήσει ένα μητρό για την καταγραφή των ιδιοκτητών και δικαιούχων, όμως δεν υπάρχουν εγγυήσει και δεσμεύσεις για τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο μητρό. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναθεωρήσουμε την ομοθεσία για το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο διεθνής έλεγχος και η εποπτεία των τραπεζών. Η εσθονική θηγατρική της Danske και έχει καταδικαστεί για φορολογικές απάτες μετά από την υπόθεση Μανίτσκι το 2008. Χρησιμοποιήθηκε και στο λεγόμενο Landromat της Ρωσίας, το ρωσικό Landromat, υπήρξε μια έκθεση που δείχνει ότι 20 δις δόθηκαν εκτός Ρωσίας από επιχειρήσεις στη Μολδαβία και σε άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή πήγαν στην Λετωνία τα χρήματα αυτά, κινήθηκαν σε πάρα πολλές άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από ε, δεκάδες χιλιάδες μάλλον συναλλαγές έγιναν μέσω των ευρωπαϊκών αυτών τραπεζών και δεν παρενέβησαν κεντρικές αρχές ή και κεντρικές τράπεζες όπως και στην περίπτωση της Εσθονίας. Τα email για τις συναλλαγές αυτές δείχνουν ότι η εσθονική εποπτική αρχή ανησυχούσε για τους Ρώσους πολίτες που ήταν πελάτες των εσθονικών τραπεζών και ταυτόχρονα ήρθαν σε επαφή με την Danske Bank και ανησύχησαν γιατί η Danske δεν αντιμετώπιζε το θέμα αυτό σοβαρά. Οι διεθνείς νομικές ρυθμίσεις ε, δεν έχουν πολλά μέσα για να επιβάλλουν κυρώσεις ε, σε νομικά πρόσωπα, αλλά παρόλα αυτά οι αρμόδιες αρχές, οι τα κτλ. θα πρέπει να αναλάβουν δράση σαν παράδειγμα απόσυρση ε, της άδειας λειτουργίας πιστοτικών ιδρυμάτων που συστηματικά παρανομούν. Στην Λετωνία με μετά την υπόθεση Μανίτσκι έξι, έξι τράπεζες μεγάλες ε, φάνηκε ότι εμπλέκονται. Ε, μία από τις τράπεζες αυτές έπαιζε σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ρωσικού Λαντρομάτ και το Μάρτιο του 16 της απεσήρθη η άδεια λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για συστηματικές και σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας για το πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μεγάλες τράπεζες λειτουργούν μόνο γι' αυτό. Είναι πολύ εύκολο να είναι κανείς ιδιοκτήτης μιας τράπεζας όταν καλύπτονται οι ανάγκες που έχει για το ύψος των συναλλαγών κτλ και νομίζω ότι έχουν υπάρξει αντίστοιχα τέτοια σκάνδαλα και στη Βραζιλία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι υπήρξε πραγματική ουσιαστική εποπτεία για τον έλεγχο των συναλλαγών αυτών. Παρακολουθούσαν πραγματικά το τι συνέβαινε στις τράπεζες αυτές τις οποίες πολλές φορές είχαν υψηλό επίπεδο συμμετοχής. Έχουν ξεκινήσει βέβαια τον τελευταίο καιρό κάποιες έρευνες, αλλά πάρα πολλές από τις υποθέσεις δυστυχώς δεν έχουν πάρει ακόμα απαντήσεις. Εμείς το Transparency International Έχουμε πάρα πολλά, θα έλεγα, συμπεράσματα βγάλει από τις υποθέσεις αυτές. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια του δημοσίου μητρώου δικαιούχων και ε, καταθετών και έλεγχος φυσικά των δηλώσεων συμμετοχής και υποχρεωτικός φυσικά χαρακτήρας συμμετοχής. Έλεγχος επίσης των κυρώσεων που επιβάλλονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περίπτωση που δεν υπάρχουν έλεγχοι από πλευράς τραπεζών ε, των πελατών τους. Οι, υπεύθυνοι, οι υπεύθυνες εισαγγελικέ αρχές ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα με τις τράπεζες και σε επίπεδο νομικών προσώπων και σε επίπεδο προσώπων φυσικών δεν θα πρέπει να έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο κυρώσεις και διαδικασίες αστικού τύπου αλλά και ποινικού τύπου και έχουν ξεκινήσει ευτυχώς στην Ολλανδία κάποιες διαδικασίες όπου η ING είναι σε διαδικασία ελέγχου για ποινικέ ευθύνε ε, σε συναλλαγές τις οποίες έχει προχωρήσει. Θα πρέπει επίσης οι αρμόδιες αρχές να δημοσιεύουν το ταχύτερο δυνατόν στοιχεία ενημέρωσης για τις δραστηριότητές τους και θα πρέπει να ενημερώνεται επίσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται τα μέτρα καταπολέμησης βρώμικου χρήματος ανά χώρα. Είναι κάποιες παρατηρήσεις, συστάσεις αν θέλετε. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ντόλαν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συστάσεις και αυτό που μου προκάλεσε μεγαλύτερο σοκ είναι αυτή η εικόνα η οποία παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι. Το το θέμα του, της ιδιοκτησίας θα πρέπει κατεπηγόντως να επιληθεί στην έκθεσή μας, γιατί αυτό προφανώς έχει να κάνει και αυτά που ζήσαμε στην περίπτωση των εγγράφων του Παναμά για πλαστές διευθύνσεις οι οποίες ε, εμφανίζονται σε... μαζικά. Δεν θα ήθελα όμως να σχολιάσω τις δύο παρεμβάσεις, ε, παρά να δώσω παρά αυτά το λόγο στους δύο συνεισηγητές. Ο κ. Κόφουτ είναι ο πρώτος που στον πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις δανούς δημοσιογράφους και την διεθνή διαφάνεια, την Transparency International που βρίσκεται εδώ πέρα μαζί μας. Μία πρώτη ερώτηση προ του δημοσιογράφου. Είπατε ότι αυτό που αποκαλύψατε αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα μόνο την κορυφή του παγόβουνου και θα υπάρχουν πολλά ακόμα ονόματα άτομα αποδοχής των χρήματων αυτών που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Αυτό νομίζω από μόνο του καταδεικνύει ότι είμαστε μάρτυρες σε μια διεφθαρμένης ελίτ πολιτικών σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη δικτατορία του Αζερβαϊτζάν για να συνθέσετε την εικόνα μιας ε, χώρας που είναι αντίθετη με την πραγματικότητα. Σας ρωτώ λοιπόν και αναρωτιέμαι πώς ε, θα αποκαλύψουμε το πλήρες εύρος του σκανδάλου. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς από τα μεσενημέρωση, εμείς από τον πολιτικό κόσμο για να αποκαλύψουμε όλα αυτά. Δεύτερη ερώτηση προς την διεθνή διαφάνεια. Φυσικά οι συστάσεις συμπεριλαμβάνονται τι εργασίε μα τη Επιτροπή ΠΑΝΑ. Αλλά αυτό που θέλω να σα ρωτήσω είναι το εξή. Πολλέ από αυτέ τι αδιαφανεί δομέ που διαπιστώνουμε, συναλλαγέ μεταξύ τραστ, ιδρυμάτων, σε πολλαπλά επίπεδα, Μήπως μία ιδέα θα ήταν ε, οποιοδήποτε διαμεσολαβητή, οποιοδήποτε ενδιάμεσος να χρειάζεται να αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή και οικονομική δομή γιατί αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι δεν υπήρξε οικονομικός σκοπός. Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να υπάρξει ξέπλυμα χρήματος, για να, παρεμβα... να παρεμπληθούν κάποιοι άλλοι για τους διάμεσους τώρα, τράπεζες κτλ. Το είπατε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις σε ό,τι αφορά τέτοιες συμπεριφορές. Τι προτείνετε Μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Οι ΗΠΑ είναι πολύ πιο αυστηρές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε μια απροθυμία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να κινηθούμε ε, αυστηρά κατά των ενδιάμεσων. Είναι, αν θέλετε, οι διακινητέ των ναρκωτικών και οι χρήστε. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί σας ευχαριστώ. Μία πρώτη ερώτηση λοιπόν από τον κύριο Κόφωτ για τους τρεις δημοσιογράφους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καλή η ερώτησή σας και μήνες ε, περάσαμε προσπαθώντας να αποκαλύψουμε τα ονόματα αυτά και θα πρέπει να σας πούμε ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις ε, με τις offshores αυτές τις οποίες ε, τις έχουν άλλες offshores έχουμε μπλεχτεί και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά όλο και πιο πολλά κομμάτια του παζλ αποκαλύπτονται. Μία για παράδειγμα συναλλαγή προς τη Γερμανία. Κάποιοι έλαβαν τις, τα χρήματα αυτά μέσω μια εταιρεία που ονομάζεται Diamond Trade. Ο κ. Έντουαρτ Νιλίνερ, πολιτικό από τη Γερμανία που τον ε, αναφέραμε προηγουμένω ε, εμπλέκεται. Αυτό σα δείχνει πόσο δημιουργική είναι σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των χρημάτων. Η κυρία Τρέντ δεν ε, απάντησε στι ερωτησει μα Αλλά από ό,τι φαίνεται ο κ. Λίνερ είχε πολύ ενεργό ρόλο στην αποστολή χρημάτων σε Βέλγους πολιτικούς για να πληρώσει για την εκλογή του στην ε, Επιτροπή ε, Παρατηρήσης των Εκλογών στο Αζερβαϊτζάν. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε όλο και πιο πολλές τέτοιε ιστορίες να εμφανίζονται από την υπόθεση αυτή και εμείς σίγουρα θα κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Σας ευχαριστώ και έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσει αυτές για να απαντήσω κατά πόσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό οι ενδιάμεση οι τράπεζες, οι δικηγόροι να δηλώνουν τον οικονομικό σκοπό τέτοιων ε, αδιαφανών ε, δομών που δημιουργούν. Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο ήδη είναι. Πρόκειται για μια μεγάλη λοιπόν ε, κόκκινη σημαία. Δύο πράγματα θα πρέπει να κάνουν οι διάμεσοι. Είτε να εξετάζουν σοβαρά την εκάστοτε δομή για να διαπιστώνουν κατά πόσον εξυπηρετεί κάποιο οικονομικό σκοπό και κατά πόσο πρόκειται για ξέπλυμα χρήματο ή αν έχουν οποιασδήποτε ανησυχίε να προβούν σε καταγγελία για μια ύποπτη συναλλαγή. Αυτέ οι υποχρεώσει ήδη υφίστανται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δικαίωμα. Το θέμα είναι πώ εφαρμόζονται. Και είναι σαφέ από τα περιορισμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα, περιορισμένα να τονίζουν τα στατιστικά στοιχεία, ότι είναι πάρα πολύ λίγε οι αναφορέ από τον τομέα αυτό. Στη Γερμανία σε ένα χρόνο έγιναν ε, τρει ε, καταγγελίε για υποπτέ συναλλαγέ από όλο τον κλάδο στη Γερμανία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που αποτρέπει τις καταγγελίες από πλευράς των ε, ενδιάμεσων. μήπω είναι χαμηλή η ευαισθητοποίηση ή υπάρχουν προσκόμματα στο ίδιο το νομικό σύστημα. Αυτό είναι βασικό. Και μπορεί να τίθεται και θέμα κίνητρου. Και εδώ ανακύπτει και το θέμα που αναφέρεται για τις κυρώσει. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι το επίπεδο των κυρώσεων. Σε πολλέ ε, χώρε στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, ε, προβλέπονται ποινικέ διώξει και ποινικέ ε, κυρώσει σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση τη νομοθεσία στο θέμα και πάλι είναι κατά πόσο εφαρμόζονται, κατά πόσο οι εθνικές αρχές ε, κάνουν αρκετά πράγματα για να ερευνήσουν σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη Δανία. Μέσα στην Δανία διαπιστώνουμε ότι η, η αρχή επιτήρησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποτελείται από τρία άτομα. Στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις τα οποία επιτηρούν 4 άτομα προσωπικό. Είναι θέμα πόρων, ανθρωπόρων για τα άτομα αυτά που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και επίσης να προσέξουμε σε ό,τι αφορά το εποπτικό καθεστώς, γιατί είναι πάρα πολλές οι χώρες όπου η εποπτεία γίνεται από τις ίδιες επαγγελματικές οργανώσεις και ουσιαστικά δεν ε, μεταφέρουν τις καταγγελίες για υποπτές συναλλαγές προς τις αρχές και ενδεχομένως να έχει συνέπειε αυτό και για τι κυρώσει. Το επιβεβαιώνω αυτό, λέει ο πρόεδρο. Ε, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των LuxLeaks. 403 καταγγελίε. Ξεκίνησαν 67, έρευνε κατά 67 τραπεζών και τελικά μόνο μία ήταν η υπόθεση η οποία πραγματικά ερευνήθηκε. Αυτή η δυσαναλογία λοιπόν υπό το προπέτασμα της αυτο οργάνωσης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο Πίτερ Γέτσακ είναι ο επόμενος. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και τους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προσκεκλημένη είναι μια ομάδα φοιτητών της Δημοσιογραφικής ε, Σχολής της, του Σοτούρ της Γαλλίας. Please, Peter. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις αποκαλύψεις που μας κάνατε. Πραγματικά επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων ότι σε κάποια κρατημέλη υπάρχει πρόβλημα με τους δικαιούχους, τις σχετικές πληροφορίες και πώς μπορούμε να τους ελέγξουμε, να τους θεωρήσουμε αξιόπιστους. Ήθελα όμως να συγκεντρωθώ στο άλλο σκέλος, την ε, δωροδοκία Ευρωπαίων πολιτικών, κάτι που είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό. Στην διαδικασία του Λόντροματ, ε, όπως έχει ονομαστεί, υπάρχουν τουλάχιστον δύο ε, εταιρείε, ψευδοεταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναρωτιέμαι κατά πόσον υποστηρίχθηκε από τους Αζέριους στο Ηνωμένο Βασίλειο, διπλωμάτες λόγου χάρη. Ποια ήταν η διαδικασία ή πιο συνηθισμένοι. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και μετά για τα ονόματα Ευρωπαίων πολιτικών που μπορεί να εμπλακούν και στο μέλλον. Τι φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβεί. Πόσοι είναι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που θα μπορούσαν να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση αυτή βάσει των πληροφόρων που έχετε και για την ε, διεθνή διαφάνεια, την Transparency, Transparency International. Καλέσατε τις αρχές της Τσεχίας και της Γερμανίας να διερευνήσουν το ρόλο των ψεύδο εταιριών, των κούφιων εταιριών και το αν είχαν κάποια εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Εδώ λοιπόν, επειδή φαίνεται ότι προλάβαμε εδώ κάποιες αναταραχές με τον Γερμανό πρόεδρο και τον Τζέχο εισηγητή, ε, μήπως μπορείτε να μας δώσετε και άλλες καλές ιδέες. Όχι, όχι, και οι δύο θέλουμε να υπάρξει μια διευκρίνηση και μια διαλεύκανση. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα με ενδιαφέραν και τρει περιπτώσει τι οποίε αναφέρατε στη Γερμανία. Παρακαλώ, ποιο θα πάρει το λόγο για να απαντήσει, ο κύριο Μπένσεν. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Αλήθεια είναι ότι τέσσερις εταιρείε που μπλέκονται στην υπόθεση του Αζερμπαϊτζάν, η NP και η NLP, βρίσκοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο από έξω, ξέρουμε ότι υπάρχουν σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν μέσω των εταιριών αυτών. Πήγαν από το Αζερμπαϊτζάν στην Danske Bank τα χρήματα. Αλλά δεν ξέρουμε αν ε, έπαιξαν ρόλο οι διπλωμάτες. Οι εταιρείε ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχαν τους λογαριασμούς τους στην ε, ε, εστονική, στο εστονικό υποκατάστημα της Danske Bank. Τώρα για το τι αποκαλύψεις μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον και ευρωπαίους πολιτικούς. Δύσκολο να το ξέρουμε από τώρα. Είναι περίπλοκο, περίπλοκη έρευνα λόγω όλων αυτών των κούφιων εταιριών, των ψεύδο εταιριών. κρύφτηκαν στοιχεία με την παραχάραξη ονομάτων. Εάν δούμε λοιπόν όλε αυτέ τι συναλλαγέ που έχουν γίνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολο να βρούμε τι κρύβεται πίσω από τα ονόματα των εταιριών. Άνθρωποι, οργανώσεις ίσως, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε του όλες τις προεκτάσεις. Και για την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιε αποκαλύψει για ενδεχόμενη εμπλοκή Ευρωπαίων πολιτικών. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντόλεν. Ναι, δεν έχουμε επιπλέον πληροφορίες για το που, πόσο μακριά μπορεί να πηγαίνει η βαλίτσα. Βασιζόμαστε και επαφιόμαστε στου ε, στους συναδέλφους μας Τη ερευνητική δημοσιογραφία ή όσων ασχολούνται με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε κάνει την έρευνα σε σχέση με τι αποκαλύψει που έχουν γίνει ήδη δημοσίω. Παρακολουθούμε το τι έχει γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ο διεθνή μα οργανισμό έχει ζητήσει πληροφορίε Έχουμε αρχίσει συζητήσεις με εκπροσώπους της Γερμανίας από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με τη Γερμανία λοιπόν και τη Δημοκρατία της Τσεχίας βρισκόμαστε σε συνεννόηση. Αναζητούμε ε, τις αδυναμίες του τσεχικού συστήματος. Αλλά αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το θέμα τη καλής φήμη εκτός από τη σε προσόδων. Δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν θέλει εδώ να ξαπλύνει και το κακό όνομα που μπορεί να είχε πέρα από το να δώσει χρήματα. Δηλαδή υπήρχε περισσότερο μια ε, απότερη πρόθεση πίσω από όλες αυτές τις ε, Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Νταρίτ Ροζάτη από πλευρά του ΕΛΚ. Yes, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσαν. Να σας πω ότι δεν είναι σε αυτές ε, οι εμφανίσει τέτοιων ε, ποινικών αξιόπινων πράξεων στο θέμα του ξεπλήματο χρήματο. Αλλά κάθε φορά που ακούω τέτοιε υποθέσει, πραγματικά μου προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι τέτοιου είδου εγκληματικέ οργανώσει και κυκλώματα λειτουργούν στην Ευρώπη και μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά χωρί θέμα. Έχουμε δει πρακτικέ όχι μόνο για ξέπλυμα βρωμικού χρήματο, αλλά και πολιτική διαφθορά στα κορυφαία πολιτικά επίπεδα στι χώρε μα Διερωτήσει την πρώτη να την απευθύνω προς τους συναδέλφους από την ε, Δανία. Πώς είναι δυνατόν τέτοια, τέτοιος μηχανισμός ξεπλήματος χρήματος να λειτουργεί για τόσο χρονικό διάστημα. Αμέλεια. Παρανομία ή μήπως απλά παραθυράκια στην υφιστάμενη νομοθεσία οι εποπτικές αρχές. Αναφέρομαι στην Danske Bank φυσικά, γιατί οι κούφιες αυτές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στο Νομίνο Βασίλειο καταδεικνύουν ότι προφανώ το Νομίνο Βασίλειο είναι πολύ φιλικό περιβάλλον προς τέτοιες τράπεζες. Αλλά οι τράπεζες έχουν αυστηρές προδιαγραφές για την αναφορά τέτοιων συναλλαγών. Πώς ήταν δυνατόν να μην έχει εντοπιστεί, να μην έχει παρατηρηθεί το οτιδήποτε. Πώ ήταν δυνατόν να συνεχιστεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ίσως πιο πολύ προς τον κύριο Ντόλαν, αλλά και προς εσάς, εφόσον το επιθυμείτε, είσαστε ικανοποιημένοι, γιατί εξ όσου καταλαβαίνω, πλέον η υπόθεση έχει περάσει στις εθνικές αρχές από την... Ε, έχει περάσει στα χέρια της εισαγγελίας σε ό,τι αφορά και την υποπτική αρχή των τραπεζών είσαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ε, έρευνες αυτές, με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Σας αγνωμονούμε για αυτά. Είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν γρήγορα αυτές οι έρευνες ε, εντοπίζοντας τους ε, υπετίους και δίνοντας μας μια ευκαιρία να βελτιώσουμε το σύστημα ελέγχου αν θέλετε στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και στις χρηματοπιστωτικές ροές στην Ευρώπη, εντοπίζοντας τις πιο ύποπτες συναλλαγές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ο κύριος Λούντ. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Πολύ καλές ερωτήσεις και να πω και δύο λόγια γιατί κάτι που μας απασχόλησε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Danske Bank έχει παραβιάσει σοβαρά τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά την ε, έλεγχο των πληρωμών, των ροών, των ε, ύποπτων συναλλαγών. Αυτό λέμε από την αρχή, ότι υπήρξε πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Δεν υπάρχει ωστόσο οποιοδήποτε δείγμα ότι κανείς την τράπεζα πραγματικά βοήθησε ενεργά σε ό,τι αφορά δηλαδή ενεργή συμμετοχή και ενεργό ενεργή συνενοχή ατόμων στο ιστορικό της τράπεζας από δεν ήταν μόνο θέμα έλλειψης ε, εποπτείας τελικά από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια υπήρχε σε κάποιο βαθμό και ενεργός συμμετοχή και συνενοχή για την υποβοήθηση των ατόμων αυτών που κινούντουσαν ε, στα κυκλώματα αυτά. Είναι προφανώς ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι φορά την Δανέζικη τράπεζα αυτή που έχει υποκαταστήματα στην Εστονία. Φαίνεται ότι οι αρχές σε διάφορες χώρες ήταν κάπως ε, σε σύγχυση, σε καθεστώς σύγχυσης για το ποιος ήταν υπεύθυνο για την επιτήρηση του υποκαταστήματος στην Εστονία. Και προφανώς αυτή η εποπτεία δεν έγινε σωστά. Οι αρχές λοιπόν στην Εστονία θα πρέπει να εξετάσουν τις συναλλαγίες αυτές και οι σε αρχές ε, προέβησαν σε έλεγχο. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν χρειάζονταν ε, να ξεκινήσει η σωστή έρευνα γιατί δεν μπορούσαν πλέον να διαπιστώσουν τι είχε γίνει με τα χρήματα. Αυτό για το τι πραγματικά συνέβησε και ποιος ήταν υπεύθυνο γιατί και για την επιτήρηση του υποκαταστήματος στην Εστονία. Μάλιστα, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και έχετε το λόγο, κύριε Ντόλαν. Yes, Ίσως να υπήρξε πράγματι συνενοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση σε κάποιες ενέργειες. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν κάποια σάπια μήλα εδώ, είναι το σύστημα το οποίο λειτουργεί έτσι και βλέπουμε στον δίκτυ της Transparency International ότι κάποιες από τις πιο οικονομικά θα έλεγα προχωρημένες χώρες έχουν πάρα πολύ ευάλωτα συστήματα. Ε, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως η Δανία όπου ε, τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και πρωτοπόρα. Από την άλλη θα έλεγα οι Δανέζικες αρχές δεν θα πρέπει να αισθάνονται πάρα πολύ καλά όταν διαβάζουν τα ευρήματα της Task Force. Σε 36 παρατηρήσεις ε, θα έλεγα η Δανία είναι ανεπαρκής, σε κάποιες άλλες παρατηρήσεις επιμέρους μόνο. Μιλάτε για την λίστα την οποία φτιάχνετε εσείς σαν διεθνής διαφάνεια. Και μιλάμε για μία από τις πέντε καλύτερες χώρες στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις αυτές. Όπως είπα στην αρχή, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς στην Transparency International είναι ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή η διαφθορά στον δημόσιο χώρο. Στην περίπτωση των δανών δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι δωροδοκιών σε χαμηλό επίπεδο κτλ. Αλλά παρόλα αυτά η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία και στις ε, ερωτήσεις το ερωτηματολόγιο μόνο ένα τμήμα καλύπτεται ικανοποιητικά. Και από ό,τι φαίνεται ε, οι υπεύθυνοι των τραπεζών δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρος ε, στα θέματα καταπολέμησης του, του βρώμικου χρήματος και όταν υπάρχουν πρόστιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Μιλάμε για σοβαρές παρατηρήσεις οι οποίες ε, τιμωρούνται με ε, πολύ μικρά ποσά. Στο Λουξεμβούργο σαν παράδειγμα μπορεί ένα πρόστιμο για μια πολύ μεγάλη παράβαση να μην ξεπερνάει το 20-30 χιλιάδες. Ε, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες το management των τραπεζών δίνει σημασία πραγματική στο τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα. Μήπως ε, θα μπορούσε το γεγονός ότι είναι υψηλά στη λίστα σας για την ε, ε, διεθνή διαφάνεια, άλλα κομμάτια τελικά της αγοράς να εφησυχάζονται. Γιατί αν θυμάμαι καλά, στη Φιλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία και η Σιγκαπούρη είναι στις πρώτες του καταλόγου σας. Μήπως λοιπόν αυτό έχει συνέπεια. Μήπω, η Transparency International θα πρέπει να επεξεργαστεί εκ νέου τον κατάλογο αυτό. Η Άννα Γκόμε είναι η επόμενη. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου προκαλεί έκπληξη. Αντίθετα με τον συνάδελφο. Γιατί το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι σχετικά κοινό. Το είδα και στη δική μου χώρα όπου κλαπτοκράτες αγοράσαν τράπεζες από άλλες χώρες για να βγάλουν χρήματα. Ήταν σαφή τα πράγματα. Ήταν γνωστό ότι κάτι είχαν ε, τμήματα των τραπεζών και μέχρι να το καταγγείλω, κανείς δεν ενδιαφέρονταν ούτε η ΕΚΤ ούτε η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή η Εθνική Αποπτική Αρχή. Έχω ερωτήσει, κύριε Ντόλ. Είπατε ότι η πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματο όπου να είναι θα δημοσιευτεί. Αυτό δεν αληθεύει όμω πλέον, γιατί παρά το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη προωθούσαν την αναθεώρηση τη οδηγία για τι συνέπειε για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, πριν από δύο εβδομάδε, ωραία, ωραία, την μπλοκάρισαν σε ό,τι αφορούσε την διαφάνεια των καταπιστευμάτων σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις για τους ενδιάμεσους, οι golden visas, οι χρυσές αυτές θεωρήσεις, για τα άτομα τα οποία που δεν θέλουν να αποκαλύψουν τους δικαιούχους ιδιοκτήτες. Να το τονίσω λοιπόν αυτό επευκαιρίας γιατί είναι πραγματικά σκάνδαλο το γεγονός ότι το Συμβούλιο τα μπλοκάρει όλα αυτά αφότου το Κοινοβούλιο ολοκληρώσε τις δικές του, το δικό του τμήμα των εργασιών. Ερώτημα λοιπόν. Αυτό που μας αποκαλύπτεται είναι ότι είναι η ίδια δημοκρατία η οποία τελικά διακυβεύεται και απειλείται. Και Οι φήμε για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο στο Αζερβαϊτζάν είχαν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξέρουμε ότι όταν πήγαμε τελευταία φορά για να παρατηρήσουμε τι εκλογέ στο Αζερβαϊτζάν μετά από το Συμβούλιο τη Ευρώπη, προβήκαμε σε μία δήλωση χωρίς να λάβουμε υπόψη τα βασικά πορίσματα του ΟΝΤΙΡ κτλ. Αυτό τότε λοιπόν προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο στην Ευρώπη και να αναρωτιέμαι κατά πόσον ερευνήσατε αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά πόσον συμμετείχαν. Θυμάμαι ο κύριος Αρλάκης, ο οποίος πλέον δεν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία άλλη ερώτηση σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τη Μάλτα. που προέκυψε με τη δολοφονία της κυρίας Δάφνη Γαρουάνα Γκαλίσια στα προγράμματα επενδυτών όπως αναφέρονταν. Έχετε στοιχεία, ξέρετε τίποτα για τη σύνδεση αυτή ενδεχομένως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Πράγματι συνειδητοποιούμε όταν αρχίσαμε να εξετάζουμε την υπόθεση αυτή συλλέξαμε στοιχεία και πρόσωπα τα οποία θα έλεγα δεν ακολουθούσαν τον γενικό κανόνα σε σχέση με το Αζερβαϊτζάν. Αυτοί στους οποίους έχουμε αναφερθεί είναι αυτοί οι οποίοι τεκμηριωμένα έχουν πάρει χρήματα. Αυτό είναι ο ρόλος μας ως δημοσιογράφοι. Για την περίπτωση της Μάλτα, στην οποία αναφερθήκατε, πράγματι προσπαθήσαμε, όπως είπε και η συνάδελφος, να δούμε αν υπάρχουν παράλληλες εξελίξεις ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχουν ονόματα εταιριών, τραπεζών, πολιτικών, δικαιούχων δεν υπάρχουν προφανείς ομοιότητες ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Η περίπτωση της Μάλτας εμπλέκει τράπεζες από το Ντουμπάι και και ε, επίσης επιχειρήσεις στον Παναμά ιδιοκτησίας Ντουμπάι που φτάνουν ίσως σε κάποιους πολιτικούς στη Μάλτα. Αντίστοιχο με την υπόθεση της Ντάνσκε στην Εστονία αλλά παρόλα αυτά οι περιπτώσεις μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν βλέπουμε κάποια κοινότητα πρωταγωνιστών. Το θέμα είναι αν συνεχίσουν να υπάρχουν ε, αυτά τα, δύο, αυτά τα λάνδρομα, τότε αυτές οι δύο περιπτώσεις μπορεί να μας βοηθήσουν να δούμε στο μέλλον πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το όνομα της είναι τη συζύγου του Πρωθυπουργού τη Μάλτα εμφανίζεται στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριο ε, Όρμπαν από την ΚΟΕ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, Δανούς δημοσιογράφους να μου μιλήσουν για τη διπλωματία του ε, στο Χαβιάρι, με Χαβιάρι και να αναφερθώ στον Πέδρο Αβραμόν. Ο Πέδρο Αγραμούν ήταν πρόεδρος του κοινοβουλευτικού, ε, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβολίου της Ευρώπης μέχρι τον Οκτώβριο. Παρετήθηκε ε, αυτός ο γερουσιαστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος γιατί διάφορα μέσα ενημέρωσης τον ενέπλεξαν με άμεσο τρόπο στη στην διπλωματία του Χαβιαριού. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε σε ονόματα και υπάρχουν πολλοί περισσότερα, εσείς τι πιστεύετε για την εμπλοκή του Πέδρο Αγραμούν στην λεγόμενη αυτή τη μορφή της διπλωματίας με το Χαβιάρι. Είπαμε παρετήθηκε από την Προεδρία της συνέλευσης του Συμβουλίου αλλά παραμένει γερουσιαστής στη Μαδρίτη. Και θα ήθελα να μην παραμείνουμε μόνο σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Ντόλαν για το Αζερβαϊτζάν που είναι σημαντικά αλλά τα εξαντλήσαμε εν μέρη και να μιλήσουμε λίγο για το μητρό των τελικών δικαιούχων. Ένα μητρό το οποίο οφείλει να είναι αξιόπιστο και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα των εργασιών μας πρέπει να πούμε ότι τίθεται και επίσης τίθεται επίσης το θέμα των κυρώσεων. Ε, αποτρεπτικές πρέπει να είναι οι κυρώσεις αυτές σε σχέση με τους ενδιαμέσους, τους διαμεσολαβητές. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στην φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ Μιγγέλ. Ο κύριος Λούντ. Ευχαριστώ. Ναι, γνωρίζουμε την περίπτωση Έγκραμοντ και τις σχετικές εκθέσεις της διπλωματίας Έχουμε ελέγξει όλε τι συναλλαγές που πήγαν σε ισπανικέ εταιρείε και ισπανού δικαιούχου. Δεν εμφανίστηκαν όμω ονόματα πολιτικών ε, από τι δικέ μα δουλειά, από τα δικά μα στοιχεία. Το χρήμα πήγαινε σε εταιρείε που λόγω χάρη πολλούσαν υλικό για κατασκευαστικές στην Ισπανία ή είδη πολυτελεία επίση στην Ισπανία, αλλά δεν υπήρχαν ονόματα πολιτικών. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση τη Κάρεν Στρίντς τα χρήματα πήγαν μέσω άλλων, τρίτων σε αυτήν. Δεν θέλω να αποφανθώ εδώ, απλώς ε, να επαναλάβω ένα από αυτά που είχαμε πει και προηγουμένως. Δεν μπορούμε να δούμε τους δικαιούχους αυτών των ε, offshore εταιριών. Μπορεί να βρίσκονται και ενδιαφέροντα ονόματα πίσω από αυτά. Δεν λέω ότι είναι από αυτούς ο Άγκραμον, αλλά Μπορεί απλώ να βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου, Απλώ δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε εδώ. Πρόεδρε, μια ερώτηση μόνο. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις, έχετε να αναφερθείτε σε κάποιες ε, συγκεκριμένες, ε, στην περίπτωση της Βαλένθια, σαν παράδειγμα έχετε κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι αν υπάρχουν κάποιε στη Βαλένσια, μπορώ όμω να ψάξω και να σα ενημερώσουμε. Θα το ελέγξουμε. Σα ευχαριστώ. Κύριε Ντόλαντ. Ευχαριστώ. Νομίζω μπορώ να είμαι σύντομος. Μιλήσατε για μητρό καταγραφή των δικαιούχων. Όμω τα στοιχεία πρέπει να μπορούμε να τα επαληθεύουμε και να τα ελέγχουμε. Κυρώσει. Θα επαναληφθώ. Προφανώ δεν ε, λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι πολύ χαμηλά τα πρόστιμα. Και σχεδόν είναι λες και κάνουμε ε, ντά τις εταιρείε που κάνουν κάτι το παράνομο. Αυτό που θα έχει σημασία είναι οι senior manager των τραπεζών να ε, προσαχθούν ε, για εγκληματική δράση. Αυτό έχει ήδη προταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για το σύστημα των senior manager. Αυτό θα ήταν ένα καλό μοντέλο. Και μετά ο ρόλος των επαγγελματικών φορέων και ενώσεων σε όλα αυτά. Ακούσαμε ότι η διάμεση είναι εμπόριο ναρκωτικών πολλές φορές. Όλοι γνωρίζουν ε, τις επιπτώσεις των, ε, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, της νομιμοποίησης. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να τις αναλαμβάνουν. Γιατί να μην χάνουν οι λογιστές και οι δικηγόροι τις επαγγελματικές τους άδειες. Αυτό θα ήταν μια τιμωρία. Εγώ δεν έχω δει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν έχουν χάσει την δυνατότητα να ασκούν την επαγγελματική του δραστηριότητα ω τιμωρία. Φυσικά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν μορμένες υποθέσεις, αλλά ε, δεν ε, συγκρίνονται με τα μεγαλύτερα αυτά φαινόμενα. Ο κύριος Σούλα από τους Πράσινους έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τον Οκτώβριο υπέβαλα μία τροπολογία για την ε, έκθεση της Ολομέλειας για την διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που καλούσε το Κοινοβούλιο μας ε, να ξεκινήσει συνεκτική και ευρεία έρευνα ε, σε ό,τι αφορά τέτοιες σχέσεις και τη σχέση με άλλα αυτορχικά καθεστώτα. Αυτή η τροπολογία συνυπογράφηκε από δεκάδες βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα Χαίρομαι που σήμερα λοιπόν συζητάμε τις υποθέσεις αυτές στην Επιτροπή Πάνα και νομίζω ότι είναι σαφή η σύνδεση μεταξύ του ξεπλήματος χρήματος από αυταρχικά καθεστώτα και το πώς προσπαθούν να επηρεάσουν τους πολιτικούς και τους πολιτικούς ευθύνοντες για να αυξηθεί η επιρροή τους στις χώρες σε ό,τι αφορά την άμεση σχέση μεταξύ των ψευδών παρατηρητικών επιστολών και των ε, υπεύθυνων από την Αζερβαϊτζάν, όπως είπε και η Άννα Γκόμες, ε, διάφοροι πολιτικοί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία και το καθεξής, ε, κατηγορούνται για δωροδοκία για συμμετοχή σε αποστολές στο Αζεμπάιτζαν προέβησαν σε θετικές δηλώσεις μετά τις εκλογές στο Αζερβαϊτζάν. Και όπως είπατε, περιλαμβάνονται και μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση αυτή. Ωστόσο, φοβάμαι ότι στην δημόσια ακρόαση αυτή, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και απαραίτητη, δεν ε, θα την καταστήσει, αντικαταστήσει την ε, ανάγκη του Κοινοβούλου να συστήσει ειδική ερευνητική επιτροπή γιατί αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε πρόσκομα προς τα καθεστώτα αυτά που συνεχίζουν να διαφθείρουν. Ναι, και κλείνω στο σημείο αυτό, Πρόεδρε. Να σας πω ότι το εταιρικό αυτό οικοδόμημα έχει ε, επανειλημμένα εξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Οι σχέσεις με τα αυταρχικά καθεστώτα πάντα παραβλέπονται. Έχετε λοιπόν συστάσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ σημαντική και δυνάμει καταλητική πηγή διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, και θα πρέπει να προσέξουμε την ώρα, γιατί αργήσαμε να καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο. Τι συστάσεις έχετε να κάνετε προς το Κοινοβούλιο, προς τους βουλευτές που που λοιπόν, αν θέλετε, εγκάρσια ατομή εκπροσώπησης των πολιτών ε, από το πολιτικό, οικονομικό κόσμο κτλ. Έχετε το λόγο για συστάσεις. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, κ. Μπέντσεν. Yeah, thank you for your, for your question. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να δώσουμε μια σαφή πολιτική σύσταση εδώ. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι, ε, που μπορούμε να εντοπίσουμε από μια τέτοια υπόθεση είναι το τεράστια ομάδα τέτοιων εταιριών που ως τρόση καλύπτουν ε, με τα slash fund ε, δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι δύσκολο να ερευνηθούν τέτοιες υποθέσεις και να βρούμε τους πραγματικούς δράστες. Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίσαμε στην έρευνα αυτή ήταν ένα θέμα δικαιοδοσίας. Είναι τεράστια η Δανέζικη Τράπεζα που ε, ε, είναι αντικείμενο εποπτεία από τι Δανέζικε Αρχέ στην Κοπενχάγη, μεν, αλλά το υποκατάστημα τη Εστονία, το... τη θηγατρική τη Εστονία την ε, εποπτεύει η Εστονική Αρχή. Είναι δύσκολο λοιπόν οι αρχές ε, της Κοπεχάγης και του Τάλιν να συντονιστούν και είναι και δύσκολο να καθορίσει κανείς ποιος ερευνά τι και ποιος εποπτεύει τι. Αυτό κάπου χάνεται στην πορεία μεταξύ της Δανίας και της Εστονίας. Είναι ε, λίγο μπερδεμένο το τι πρέπει να ερευνήσει κάθε αρχή για όλες τις αρχές. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια θέματα, θέματα δικαιοδοσίας. Κύριε Ντόλαντ, ευχαριστώ. Γνωρίζω την υπόθεση του Ευρωκοινοβουλίου που επενηχθήκατε και εσείς, προτίσατε και εσείς ο Πρόεδρος. Δεν είναι το επίκεντρο των κατηγοριών το Κοινοβουλίο. Το κάθε Κοινοβούλιο οφείλει να προσπίσει τον εαυτό του από τέτοιου είδου παράνομε δραστηριότητε και να προστατεύει την ακεραιότητά του. Αλλά αυτό που είδαμε σε όλη την Ευρώπη είναι ότι, όπω και στην περίπτωση των ε, μεσαζόντων, θα πρέπει κάπου να υπάρχει λογοδοσία και επιβολή κυρώσεων. Αυτό ισχύει και για του βουλευτέ και για του μάνατζερ των τραπεζών. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει είναι η τάση που έχει ξεκινήσει στη Γαλλία και αλλού στην Ευρώπη να υιοθετηθεί γενικότερα. Ε, ανεξάρτητοι φορεί να ερευνούν τα θέματα αυτά και την ακαιρεότητα και την ανεξαρτησία των βουλευτών να μπορούν έτσι να την προστατεύσουν. Θα προτείναμε στου ευρωβουλευτέ να κοιτάξουν και αυτή την αναλλακτική. Για μια τελευταία παρατήρηση ίσω να πω ότι αυτό θα λαμβάνει λίγο και μεγαλύτερη σημασία, διότι γνωρίζουμε από αυτές τις αλλά και αποκαλύψει αλλού ότι οι αντιδημοκρατικοί θεσμοί δέχονται Μάλλον ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται διαρκώ συστηματικέ επιθέσει από άλλε κυβερνήσει που προσπαθούν να τι υπονομεύσουν. Η εμπιστοσύνη μου στι ε, δυνατότητε αυτοκάταρξη, αν θέλετε, των δημοκρατικών καθεστώτων δεν έχει ακόμα διαψευστεί. Και θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν προκειμένου οι ομάδε φιλία να βοηθούν, γιατί οι ομάδες φιλίε συνήθω ε, χρηματοδοτούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσει αντίθετα με τι ε, ομάδες αποστολών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το τονίζω σε ε, όταν μιλάμε για ομάδες φιλία. Μάλιστα, ο κύριο και τέλος ο Ντάριος Ροζάτη, αν έχει και αυτό μια ερώτηση να κάνει. Ντέιβιτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως βλέπετε, και όπως είπατε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χαμηλό κόστος για την έναξη εταιρεία. 12 α, 12 λίρες. Γιατί, όχι, στην Ηνωμένο Βασίλειο το ονομάζουμε στο δημοκρατικό καπιταλισμό. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ξεκινήσουν μια εταιρεία. Ανεξάρτητα από το πόσο χρήματα έχουν να διαθέσουν. Όσο και λίγα να έχουν να διαθέσουν. Και αυτό θεωρώ οδηγεί σε μια δημοκρατική και δυναμική οικονομία. Πιο πολλέ θέσει εργασίας. Κάποιοι γελούν. Α, κάποιοι από αυτού που έχουν ε, τελείω ε, σάπιες οικονομίε και μεγαλύτερη ενεργία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όσο πιο πολύ περιπλέκονται τα πράγματα, τόσο πιο πολύ αποτρέπουμε τον κοσμάκι από το να συστήσει μια εταιρεία. Και γι' αυτό όλο και πιο πολλές κόσμος ε, ζει τελικά και από το του κράτος. Αυτό θέλετε να κάνετε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και εξηγεί γιατί η Γαλλία είναι λιγότερο δημοκρατική και γιατί ο κόσμος έχει λιγότερη ευημερία. Γιατί δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με το κράτος αν θέλει να έχει μια επιχειρήση. 60% των Γάλλων ε, ζει σχεδόν άμεσα από το κράτος, όπως στο σοβιετικά κράτη. Στο σοβιετικό κράτος. Δεν είμαστε τόσο παρανοϊκοί όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά φρεχτό ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αν ε, παίρνουν χρήματα, προφανώς θα πρέπει να τιμωρηθούν. Και έχουμε ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό και δημοσιογραφικό μηχανισμό που τα φροντίζει αυτά. Ναι, έχετε δύο λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι δήλωση, είναι απαντώ σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, γιατί μιλάνε για τις επιχειρήσεις. Κάποιος θα πρέπει να υποστηρίξει σε αυτό το κτίριο της ε, εταιρείας. Ευχαριστώ για τη δήλωση, δεν χρειάζεται απάντηση στις δηλώσεις. Ε. Νταρίς Ροζάτη. Όχι παραπάνω, γιατί θέλω να δώσω και στους δύο ομάδες ομιλητών ε, ένα λεπτό για να απαντήσουν και να συνοψίσουν. Κύριε Ντόλαν. First Πρόεδρε, να πω και εγώ ότι θεωρώ ότι αυτά που ακούσαμε σήμερα από τους δημοσιογράφους ε, δείχνουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη όλα. Και επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τέτοια συστήματα λόντρωμα πλυντηρίου ε, που Πρέπει να τα παρακολουθήσουμε στενά, να τα ε, φέρουμε στο φω, να κοιτάξουμε όλε αυτέ τι υποθέσει και θα το κάνουμε με το ποιο τρόπο μπορούμε στην Επιτροπή μα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υποθεί. Επίση, να πω ε, ότι λυπάμαι κύριε Κόμπερν για τα σχόλια σα, αλλά αυτό που μα λέτε είναι ότι κάθε πολίτης να έχει έναν φορέα δικό του για να κοιτάζει τη φοροαποφυγή του. Ε, δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί να μην ήτανε. Ναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο σοβαροί εδώ. Αυτά που ακούσαμε σήμερα είναι σοβαρά. Είναι σοβαρέ περιπτώσει διαφθορά, ε, ξεπλήματο ε, χρήματο και τη καλή φήμη κάποιου, του καλού ονόματο κάποιου. Γι' αυτό λοιπόν επαφιόμαστε στου δημοσιογράφου και στην ε, Transparency International και με την αφοσίωσή μα ελπίζουμε να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Θα το κάνουμε με ποιο τρόπο μπορούμε, μόλι ξεκινήσαμε, αλλά θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ και σήμερα το πρωί συζητήσαμε στους συντονιστές το πώς θα οργανώσουμε την ε, εργασία και πώς θα συστήσουμε στο Κοινοβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε αυτό συμφωνούμε γιατί είναι μια διαδικασία ανεξέλιξη. Κύριε Ντόουλ, ε, για ένα λεπτό αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ίσως και λιγότερο από λεπτό. Τα αδύναμα σημεία του συστήματος είναι σαφή τις λύσεις μπορούμε να τις διαδούμε ε, ακόμα μόνο, αλλά είναι σημαντικό εδώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Μιλήσατε για την αναμενόμενη αναθεώρηση τη οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει εδώ το Κοινοβούλιο να βεβαιωθεί ότι κάποια από τα μέτρα που ε, το ίδιο το Κοινοβούλιο να έκρινε για την ε, προτιμησιακή ιδιοκτησία, για την ε, ενισχυμένη δέος επιμέλεια για πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όλα αυτά τα μέτρα που το ίδιο Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει να υπάρχουν στην τελική πρόταση. Για να επιβληθούν και στα κάτι μέλη και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει και να πληρώσει αυτόν τον ρόλο που του αναλογεί. Ευχαριστούμε πολύ και από εσά κάποιε απαντήσει, κυρία Λούντ. Τελικές παρατηρήσεις δεν έχω. Όποιος θέλει να μας ε, θέσει ερωτήσεις, ευχαριστώ και θα τους απαντήσουμε ε, μετά τη λήξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κηρύξω τη λήξη. Να ευχαριστήσω τους παρεμβαίνοντες. Και το γεγονό ότι δεν είχαμε πολλού συναδέλφου μαζί μα στο τέλο ε, οφείλεται στο γεγονό ότι έχουμε σημαντικέ ψηφοφορίε ε, ε, στην Επιτροπή Ήτρα για το πακέτο για την ενέργεια και δυστυχώ διεξάγονται παράλληλα προ τη δική μα ακρόαση. Συνεχίζουμε λοιπόν στι 3 το απόγευμα για τα Paradise Papers. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ευγενικά ο Πρόεδρο ευχαριστεί και του διερμηνεί.